Αγαπητοί συνάδελφοι, πρέπει νομίζω να ξεκινήσουμε. Κυράει πολύ γοργά ο χρόνο, έχουμε αρκετά θέματα στην ημερήσια διάταξη για σήμερα και επίση ήθελα να σα ενημερώσω, ίσω να το θυμάστε βέβαια, γιατί το είχαμε στο ότι ε, η συνεδρίασή μα μεταδίδεται από το ίντερνετ. Έχουμε την ημερήσια διάταξη, εγκρίνεται. Ναι. Στο δεύτερο σημείο έχουμε την έκδοση των πρακτικών τη συνεδριάσεων της συνεδρίας 26 και 27 Απριλίου. Ως ήθιστε την ε, θεωρούμε ως εγκριθήσα, τα θεωρούμε ως εγκριθέντα τα πρακτικά, εφόσον μέχρι το τέλος συνεδριάσεως δεν έχουν διατυπωθεί ενστάσεις. Στο σημείο 3 της ημερήσιας διάταξης, ανακοινώσει τη Προέδρου. Ανακοινώνω ότι δεν έχω ιδιαίτερες ανακοινώσει για σήμερα και προχωρώ στο σημείο 4 για να σας ενημερώσω πολύ γρήγορα για τις εξελίξεις ε, σε σχέση με τις εργασίες ομάδας εργασίας για το μέλλον της πολιτικής συνοχής. την προηγούμενη φορά, αλλά και σε κάθε μας συνεδρίο ουσιαστικά συζητήσαμε τα θέματα τα σχετικά με το μέλλον της πολιτικής της συνοχής και πρόσφατα μάλιστα συζητήσαμε και την δομή και πράγματα που θα έπρεπε να μπουν στην, ε, στις προτάσεις μας. Οι, ομάδες, οι πολιτικές ομάδες επίσης ε, διατύπωσαν τις απόψεις τους, τα κύρια θέματα που αφορούν την πολιτική της συνοχής. Και έτσι έχουμε ένα έγγραφο εργασίας ως βάση εργασιών από την προηγούμενη μας ε, συνεδρίαση. Επίσης, επί τη βάση των συζητήσεών μας και βέβαια και των ε, πολιτικών ομάδων, ετοίμασε η Γραμματεία ένα σχέδιο εγγράφου θέσεων που θα συζητήσει αύριο η ομάδα εργασία και επίσης στόχος μας είναι η ανταλλαγή απόψεων να ολοκληρώσει τις θέσεις το ταχύτερο δυνατό μετά την αυριανή συζήτηση έτσι ώστε αυτές μετά να πάνε στα μέλη της ομάδας εργασίας, της Επιτροπής μάλλον, για να γίνει η ανταλλαγή απόψεων και να εγκριθεί από την πλειοψηφία μας το σύνολο αυτών των προτάσεων πριν από το τέλος Ιουνίου, στη τελευταία μας συνεδρίαση. Και αν εξασφαλίσουμε την πλειοψηφία βέβαια, το έγγραφο μαζί με τη συνοδευτική επιστολή της Προέδρου θα πάει και στον Πρόεδρο βέβαια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, αλλά και πρώτα απ' όλα στον, στον πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, στον αρμόδιο επίτροπο για την περιφερειακή πολιτική και όλα τα αρμόδια και εμπλεκόμενα όργανα που από κοινού ή άλλως θα ορίσουμε. Αυτά το Έχουμε αύριο από Έχουμε και επίσκεψη αύριο από, την, από συναδέλφους ε, της Ρέτζη. Θα ήθελα να δώσω το λόγο τώρα στον Μάρκος Πίβερ. Κύριε Πίπερ, χωρίς μικρόφωνο, δεν ακούγεται. Δεν ακούγεται το μικρόφωνο του κύριου Πίπερ. Ναι, ε, έχουμε και την συναγωνισμό με τους σοσιαλιστές, με συγχωρείτε τους σοσιαλδημοκράτες. Λοιπόν, το έγγραφο αυτό της ομάδας εργασίας το είδαμε. Ξέρετε ότι η πολιτική μου ομάδα έχει υπόψη πως έχω εξαρχίσει την εντυπώση της επιφυλάξης μου. Οι προτάσεις συγκεκριμενοποιούνται σιγά σιγά, κατά την άποψή μου συγκεκριμενοποιούνται υπερβολικά και νομίζω ότι εάν προχωρήσουμε στην τωρινή φάση με τόσο συγκεκριμένες θέσεις, χάνουμε πολλές ευκαιρίες. Νομίζω ότι θα ήταν καλό να είμαστε πιο ελαστικοί. Ναι, να είναι ομάδα εργασία, αλλά όχι να προσδιορίσει το μέλλον με τι εργασίε τη της πολιτική τη συνοχή. Αυτό είναι κάτι το οποίο δεν μπορεί να γίνει τώρα γιατί δεν έχει προχωρήσει επαρκώ ο διάλογο. Δεν είναι όριμο και γι' αυτό θα ήθελα να είμαστε πολύ προσεκτικοί ω προ το συγκεκριμένο έγγραφο εργασία. Η πρόεδρο, ευχαριστώ. κοιτάξτε, του άλλου. Εμεί θα κρίνουμε πόσο δεσμευτικέ θα να είναι οι αποφάσει, δεν υπάρχει ω προ αυτό αμφιβολία. Η κυρία Σρότερ, θα ήθελα και εγώ να επισημάνω ότι εξ αρχή είχα εκφράσει την ε, υποστήριξη μου σε αυτέ τι επιφυλάξει του συναδέλφου κυρίου Πίπερ και στην ομάδα εργασία και στου συντονιστέ. Επαναλαμβάνουμε διαρκώ ότι η διαδικασία αυτή σε επίπεδο Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου θα πρέπει να αφορά του κύριου πυλώνε μια ε, της μεταρρύθμισης ε, πολιτικής της συνοχής, ότι χρειάζεται επαρκή χρόνο, επαρκή διάλογο αυτή η διαδικασία, επαφή και επικοινωνία με τις διάφορες περιφέρειες και λήψη υπόψη των διαφορετικών του συνθήκων και χαρακτηριστικών. Και νομίζω ότι αυτό δεν το έχει επιτύχει η ομάδα ε, εργασίας υψηλού επίπεδου. Καλό είναι βεβαίως οι ομάδες να κάνουν τη διερευνητική δουλειά βεβαίως, συγκεκριμένη διερευνητική δουλειά που έχει γίνει, μάλιστα ορισμένε ομάδε ξεκίνησαν αρκετά ε, έγκαιρα και περιορίστηκαν σε μια γενική μόνο εξέταση της κατάστασης. Κάποιες άλλες κοίταξαν και τη γενική, αλλά και τα, τη γενική κατάσταση, αλλά και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Εν πάση περιπτώσει όμως, όπως έχω πει και ήδη στο παρελθόν, αυτό που βλέπουμε τώρα ως πρόταση δεν είναι, ως πρόταση γραμματείας, δεν είναι η σύνοψη των όσων έχουμε συζητήσει. Είναι μία μονομερή θεώρηση της κατάστασης. Φυσικά δεν μπορούμε να απαιτούμε από τη γραμματεία να προβαίνει σε εξισορρόπηση πολιτικών θέσεων. Μόνο απόπειρα εξισορρόπηση θα μπορούσε να ε, περιμένουμε, μπορούσαμε να περιμένουμε από τη γραμματεία. Εν πάση περιπτώσει όμως νομίζω ότι καλό θα ήταν να επισημάνουμε ότι υπάρχουν πολλά πράγματα τα οποία δεν λαμβάνονται υπόψη, ότι υπάρχουν αντιφάσεις σε πολλά ζητήματα μεταξύ μας, αντιθέσεις και δεν έχουμε καταλήξει συνένεση σε πολλά από τα σημεία. Υπάρχουν αντιπαραθέσεις απόψεων, διαφωνίες, όλα αυτά δεν τα καταγράφει το έγγραφο. Ή μη τι άλλο δεν καταγράφει ότι υπάρχουν διαφορετικές απόψεις. Ούτε καν αυτό. Και νομίζω ότι ιδιαίτερα σημεία ενδιαφέροντος για την κάθε πολιτική ομάδα πάλι δεν καταγράφονται επαρκώς. Το ίδιο βλέπω οπωσδήποτε για την δική μου πολιτική ομάδα αλλά και για τους αλληδημοκράτες και για τους φιλελευθέρους και για τους ε, συντηρητικούς. Το ακούω πάντοτε από τις τοποθετήσεις των συναδέλφων ότι δεν έχουν εκφραστεί οι θέσεις τους μέσα στο έγγραφο και νομίζω ότι θα πρέπει να καταστήσουμε σαφή αυτή την κατάσταση, να την καταγράψουμε και να δούμε ποιο είναι το σημείο στο οποίο συναντιούνται οι διαφορετικές μας απόψεις. Δεν μπορούμε όλα αυτά όμως να τα κάνουμε μία ένα συνονθήλευμα και να λέμε ότι βγαίνει από εκεί η ουσία. Ξέρω ότι είναι μια δύσκολη πολιτική ε, διαδικασία, ξέρω όμως ότι δεν την έχει επιτελέσει αυτή η δουλειά η γραμματεία. Αυτή τη στιγμή λοιπόν καλό θα είναι να έχουμε διαρθρωμένες συζητήσεις μέσα στην Επιτροπή να εκφράζουμε τις θέσεις μας, να μπορούμε να, εκφράζει, να μπορεί να ο καθένας να εκφράζει τις θέσεις του και από εκεί και πέρα να προκύπτουν οι θέσεις πλειοψηφίας, ενδεχομένως της μειοψηφίας να καταγράφονται ή παραδείγματι να καταγράφεται στο έγγραφο ότι εδώ διαφοροποιήθηκαν κάποιες ομάδες ή κάποιοι βουλευτές και από εκεί και πέρα να είναι σε θέση και το Κοινοβούλιο ολόκληρο να αποφασίσει τα περαιτέρω. Οπότε δεν υπήρξε στο θέμα αυτό ενότητα πνεύματος, συνένεση στην ομάδα μας και στο Κοινοβούλιο γενικότερα και δεν μπορούμε τώρα να περιμένουμε ότι αυτό θα εκφραστεί ξαφνικά στην, στο έγγραφο της ομάδας εργασίας. Κύριος Φωνίστηλ. Λοιπόν. Ευχαριστώ πολύ. Αυτή η διαδικασία να βγουν οι προσανατολισμοί σε μια πρόορη φάση είναι πειραματική διαδικασία. είναι φυσιολογικό να ξεφεύγει λίγο από το φυσιολογικό. Αυτό είναι, ο... Αυτό είναι το αντικείμενο εξάλλου. Αυτό είναι ο στόχος. Τι θέλουμε. Θέλουμε να ενισχύσουμε την πολιτική συνοχή. Και αντί να μιλάμε διαφορές, καλύτερα να επιμένουμε στη συνοχή. Κρίμα που Σύντομα θα μιλήσουμε για τη χρηματοδότηση. Όλοι ασχολούνται με αυτό, όλοι παραπονιόνται για το ότι δεν, υπάρχουν, δεν υπάρχει έγγραφο. Εγώ το βλέπω λίγο διαφορετικά το θέμα. Πιστεύω ότι μπορούμε να ψηφίσουμε για το έγγραφο αυτό. Μπορούμε να καταθέσουμε τροπολογίες αν το θέλουν οι συνάδελφοι αλλά είναι μια ενδιάμεση φάση. σε σχέση με τη μελλοντική χρηματοδότηση. Πρέπει να κάνω μια πρόταση με το κείμενο αυτό. Μπορούμε να το αποκαλέσουμε και έκθεση το έγγραφο αυτό και να καταταθούν τροπολογίες. Υπάρχουν διαφορετικές απόψεις, το είδαμε αυτό στην Ολομέλεια. Η χρηματοπιστωτική κρίση είναι ένα εμπόδιο για τη συνοχή. Αν ο κύριος Πίπερ θεωρεί ότι το κείμενο είναι υπερβολικά λεπτομεριακό, ας προτείνει τροπολογίες διαγραφής. Η συζήτηση έχει ξεκινήσει. Μερικοί θέλουν η συνοχή να είναι πολύ ασθενής και να υπάρχουν ε, προϋπολογισμοί κατά τομέα. Αυτός δεν είναι ο δικός μας στόχος. Εμείς θέλουμε να κάνουμε μια έκθεση στην ομάδα εργασίας. Ας καταθέσουμε λοιπόν τροπολογίες σαν να ήταν έκθεση. Κύριε Πρόεδρε, νομίζω ότι θα πρέπει να υπενθυμίσουμε τι είχαμε επιδιώξει με το έγγραφο αυτό. Με το έγγραφο λοιπόν προσπαθήσαμε, θελήσαμε να προετοιμάσουμε μια πολύ σημαντική συζήτηση, την οποία έπρεπε να κρίνει το Κοινοβούλιο επιτέλους και δεν νομίζω ότι είναι η πρώτη φορά που το με αυτό πολλούς. Ε, μια συζήτηση λοιπόν η οποία πάντοτε ήταν πολύ περίπλοκη, που πολλές φορές χρειάστηκε να οργανωθεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και για διάφορους λόγους περιφερειακούς, εθνικούς, πολιτικούς, ή λόγους και ιδιαίτερων συμφερόντων, δηλαδή το ποιος ανήκει στην περιφερειακή, τη γεωργική ή ποια άλλη επιτροπή. Μια υπόθεση λοιπόν πολύ περίπλοκη και τελικά μετά τη συνθήκη της Λισαβόνας εφόσον έχουμε και τη δικασία της συναπόφασης για τον κανονισμό, είμαστε αναγκασμένοι να αντιμετωπίσουμε. Ιδάλλως το Κοινοβούλιο πώς θα μπορέσει να οργανωθεί πρέπει να έχει καλά επιχειρήματα, καλή συζήτηση για να μπορέσει να προχωρήσει σε μια καλή πολιτική συνοχή. Διαφορετικά θα είναι μόνο εμβαλωμετικέ οι λύσει στην πολιτική τη συνοχή. Αυτό θέλω εγώ τουλάχιστον εκ μέρου τη ομάδα μου. Αυτό πιστεύω ότι θέλουμε όλοι στην Επιτροπή μα. Θέλουμε μια καλή, συνεπή, συνεκτική προσέγγιση την οποία η Ευρωπαϊκή Ένωση θα μπορέσει να προβάλλει έτσι ώστε να προαγάγει μια αποτελεσματική πολιτική συνοχή. Εάν λοιπόν είναι αυτό που θα επιθυμούμε, μια καλή πολιτική συνοχή, τότε θα πρέπει να προχωρήσουμε βάσει αυτό το συγκεκριμένο έγγραφο θα πρέπει να το κοιτάξουμε πάρα πολύ προσεκτικά, όπως και αυτά που θα συζητήσουμε αύριο, και όντω νομίζω ότι δεν είναι σε θέση η Γραμματεία να προβεί σε πολιτικέ εκτιμήσει, ούτε καν έχει αυτό το καθήκον, την εντολή η Γραμματεία. Αλλά θεωρώ ότι δεν είναι καλή η διάρθρωση, δηλαδή δεν υπάρχει η προσέγγιση τη μεταρρύθμιση ε, τη πολιτική συνοχή μέσα στο έγγραφο. Πρόκειται απλώ για ένα άθροισμα διαφορετικών θέσεων και νομίζω ότι ανεξαρτήτω του τι θα που θα καταλήξουμε και πώς θα χειριστούμε το έγγραφο αυτό, να διαθέσουμε επαρκή χρόνο για να ξεκαθαρίσουμε τι έχει μείνει στο έγγραφο έγγραφο, τι θέλουμε να μπει μέσα στο έγγραφο, τι θέλουμε να βγει από το έγγραφο και τι λείπει από το έγγραφο και να δούμε αν μπορούμε να ταυτιστούμε η μεν και η δε με τις διάφορες θέσεις. Και αν το έγγραφο αυτό ε, μόνο για την Επιτροπή μας μπορεί να προχωρήσει κατά τον τρόπο αυτό, θα καταφέρουμε καλά. Εάν όχι, εάν βγει όπως έχει από την Επιτροπή μας, θα καταλήξουμε 300-400 διαφορετικές τροπολογίες και δεν θα μπορέσουμε ποτέ να βρούμε την άκρη. Ξεκινώ με τις μακροπεριφέρειες κάθε νήσου ανά τον κόσμο, κάθε ορεινής περιοχής ανά την Ευρωπαϊκή Ένωση, την ε, τις κυρώσεις για την ε, μη έγκαιρη καταρβολή των σχετικών ενισχύσεων κτλ. Κάθε είδους πρόβλημα θα το βρούμε μπροστά μας γιατί δεν έχει ξεκινήσει με επαρκώς συντονισμένο και διαρθρωμένο τρόπο η συζήτηση στην υπόθεση αυτή. Συμφωνώ 100% με τον κύριο Πίπερ στις παρατηρήσεις του, πρέπει να δεθέσουμε επαρκή χρόνο για τη συζήτηση. Και εν ώψη και της πέμπτης, ε, πέμπτου εγγράφου συνοχής, καλό θα είναι εμείς να είμαστε σε θέση με το έγγραφό μας να τοποθετηθούμε μέσα σε αυτές τις διαπραγματεύσεις, να έχουμε δηλαδή θέσεις για τις διαπραγματεύσεις. Είμαι πάρα πολύ επιφυλακτική λοιπόν ως προς το έγγραφο αυτό. Ευχαριστώ. Ο Ευχαριστώ. Όντως, κανένα έγγραφο δεν μπορεί να ικανοποιεί όλες τις προσδοκίες και να συμπεριλαμβάνει όλες τις απόψεις και προσεγγίσεις. Και συμφωνώ ότι θα πρέπει να προβλέψουμε και περισσότερο χρόνο. Έχω όμως μία παρατήρηση. Στη συζήτηση για την πολιτική συνοχή, πολύ συχνά υπογραμμίζουμε ότι οι προτεραιότητες αυτής της πολιτικής θα πρέπει να υπάγονται τους στόχους της στρατηγικής της ε, Ευρωπαϊκής Ένωσης για το 2020. Έχω την αίσθηση ότι στη συζήτηση αυτή πολλές φορές αμελούμε το ρόλο του πολιτισμού. Γιατί η μνήμα του πολιτισμού γίνεται πολύ ακροθυγός στην στρατηγική του 2020, μόνο επ' ευκαιρία της ανάγκης ε, ψηφιοποίησης. Θα πρέπει να αξιοποιήσουμε το δυναμικό του πολιτισμού, γιατί και το πνευματικό και διανοητικό κεφάλαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι σημαντικό για την επιχειρηματικότητα και την ευρηματικότητα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και ενισχύει την πολιτική συνοχή. Πολλοί μιλούν για την λήψη υπόψη των ιδιαιτεροτήτων των διαφόρων περιφερειών. Και μάλιστα, διαβάζοντας την έκθεση από την επίσκεψη της αντιπροσωπείας μας στην Γαλλία έχουμε την αίσθηση ότι είναι διαφορετικές οι ανάγκες των διαφόρων περιφερειών. Η κεντρική περιφέρεια της Γαλλίας δίνει έμφαση στην καινοτομία και τεχνολογική ανάπτυξη, ενώ μια άλλη περιφέρεια της Γαλλίας έχει προτεραιότητα άλλο τομέα. Μιλάει για μερικές αμέλειες που γίνονται, μερικές καθυστερήσεις, γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό στην επεξεργασία της νέας πολιτικής να διατηρήσουμε μια μεγάλη ελαστικότητα λόγω των διαφορών που υπάρχουν και των ιδιαιτεροτήτων των διαφόρων περιφερειών, ακόμη και εντός της ίδιας χώρας. Γιατί το, η προτεραιότητά μα είναι να υλοποιήσουμε τους στόχους μας. Ευχαριστώ. Δεν ξέρω αν υπάρχουν άλλα σχόλια για το θέμα αυτό. Πάντως, συνάδελφοι, όταν αποφασίσαμε για την συγκρότηση αυτής της ομάδας εργασίας, συμφωνήσαμε και για την εντολή της και για τις προσδοκίες που είχαμε από αυτή την ομάδα εργασίας. Μιλήσαμε για το πρόγραμμα της ομάδας εργασίας και το χρονοδιάγραμμα που θα εξαρτηθούν σε μεγάλο βαθμό από την ταχύτητα και το ρυθμό των εργασιών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Και αυτό θα πρέπει να ληφθεί υπόψη όταν αποφασίσουμε το θέμα της διαδικασίας και του χρονοδιαγράμματος. Και συμφωνήσαμε ότι ακόμη και με το πρώτο μας έγγραφο θέλουμε να έχουμε κάποια, κάποιο αντίκτυπο στην πέμπτη έκθεση περί συνοχής που κατά πάσα πιθανότητα θα δημοσιευθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις αρχές Νοεμβρίου και θα ολοκληρωθεί πριν τις θερινές διακοπές. Σε ό,τι αφορά τη διαδικασία πάντως, τα διαδικαστικά θέματα μπορούμε να τα συζητήσουμε με τους συντονιστές αργότερα. Δεύτερο ζήτημα είναι το περιεχόμενο του εγγράφου αυτού. Θα θυμάστε ότι είχαμε πει ότι η γραμματεία δεν ε, επεξεργάστηκε μόνο τα σχόλια της συζήτησης στην ομάδα εργασίας. Η βασική πηγή και το υλικό για τη γραμματεία ήταν τα έγγραφα που έστειλαν οι πολιτικές ομάδες. Η Πράσινη, για παράδειγμα, έστειλαν μόνο χθε τα έγγραφα αυτά. Για να μην πω και σήμερα, τελευταία στιγμή μερικέ φορέ. Και μάλιστα καμιά-δύο ομάδε δεν έστειλαν καν υλικό. Γι' αυτό ίσω οι δικέ του απόψει δεν ε, αντικατοπτρίζονται στο κείμενο. Αύριο θα γίνει συζήτηση που θα αποτελέσει και αυτή τροφή για, για τον εμπλουτισμό του, γραμ... του εγγράφου και θα περιλαμβάνει τα επίσημα σχόλια της Επιτροπής μας. Ελπίζω ότι θα καταλήξουμε σε κάτι μετά από συμφωνία για να δούμε πόσο φιλόδοξοι μπορούμε να είμαστε. Όλη αυτή την προσπάθεια συμβίλησης ε, την κάνει η γραμματεία όλων αυτών των ε, εγγράφων και του υλικού. Περιμένουμε πάντως τη συμβολή και των άλλων πολιτικών ομάδων. Τώρα, για το περιεχόμενο θα συζητήσουμε αύριο και για τη διαδικασία θα το συζητήσουμε αργότερα στους συντονιστές. Ελπίζω να έχουν προτάσεις αργότερα. Πάντως και στις συστάσεις μας για στους συντονιστές θα ασχοληθούμε με το θέμα αυτό. Αν δεν υπάρχουν άλλα σχόλια για το σημείο 4, μπορούμε να το ολοκληρώσουμε και να περάσουμε στο 5. Πραγματοποιήθηκε επίσκεψη αντιπροσωπής Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης στη Γαλλία. Επικεφαλής αντιπροσωπής αυτής ήταν ο Λαμπέρτ Βαν και μάλιστα Υπάρχει και έκθεση της αντιπροσωπείας που έχετε λάβει. Δεν ξέρω, ο Λαμπέρτη, άλλο μέλος της αντιπροσωπείας ε, που μετέβει στη Γαλλία, θα μπορούσε να μας κάνει μια σύντομη ενημέρωση για τα αποτελέσματα αυτής της επίσκεψης. Λαμπέρτη, έχεις το λόγο. Voorzitter, eh, heel graag kort en ik vraag ook de collega's waar nodig eh, er... Ευχαριστώ αγαπητοί συνάδελφοι. Ja, het is altijd een hoog tijmoment voor leden van een parlementaire commissie om, om delegatiebezoeken te brengen. Τα μέλη μιας κοινοβουλευτικής επιτροπής πάντοτε έχουν βεβαίως καλή ε, ευκαιρία να δουν τα πράγματα ε, πιο ξεκάθαρα όταν επισκέφτονται μια περιοχή. Έχουμε λοιπόν πιο καθαρή εικόνα. Αυτό ακριβώς συνέβη και με την επίσκεψη στη Γαλλία. Ήμασταν στην περιοχή της Τουρ, στην Τουρέν όπως ονομάζεται. Εκεί είδαμε τι έγινε σε σχέση με την προηγούμενη περίοδο και πόσο η πολιτική συνέβαλε στη δημιουργία των θέσεων απασχόλησης, η περιφερειακή πολιτική. Συναντήκαμε εκπροσώπους ε, τη τοπική και περιφερειακή ε, αυτοδιοίκηση και έχω την αίσθηση ότι η ενίσχυση των δομών και των δραστηριοτήτων έγιναν σε πολύ καλό περιβάλλον. Η συζήτηση στη Γαλλία είναι αρκετά περίπλοκη για το μέλλον αυτής της πολιτικής. Και σίγουρα το εργαλείο αυτό είναι πολύ σημαντικό και θα πρέπει να το διατηρήσουμε, αλλά μερικές φορές είναι δύσχριστο. Σίγουρα θα πρέπει να διδαχθούμε από τα μαθήματα του παρελθόντος. Θα πρέπει να δούμε καταρχήν αν οι στόχοι που έχουμε θέσει υλοποιήθηκαν σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο. Όλοι παραπονιούνται για την υπερβολική γραφειοκρατία που υπάρχει και ζητούν απλοποίηση των διαδικασιών και κατάργηση της υπερβολικής γραφειοκρατίας. Η γραφειοκρατία μαυρώνει κατά κάποιο τρόπο την εικόνα της Ευρώπης στα μάτια των Ευρωπαίων πολιτών. Και τα κονδύλια πηγαίνουν από τις Βρυξέλλες στο Παρίσι. Πρέπει να υπάρχει όμως ένας καλύτερος τρόπος και ευκολότερη πρόσβαση στα ευρωπαϊκά κονδύλια γιατί ο κόσμος δεν καταλαβαίνει αν πρόκειται για ευρωπαϊκά κονδύλια ή για γαλλικά κονδύλια που εκπορεύονται από την κεντρική διοίκηση, τη γαλλική. Επίσης, στις αστικές περιοχές όπως το Παρίσι μιλήσαμε για την ανανέωση των πόλεων και για την οικονομική και κοινωνική διάσταση της περιφερειακής πολιτικής. Και εκεί ακούσαμε την, το αίτημα για την υιοθέτηση μιας πιο σφαιρικής προσέγγισης, πιο ολιστικής προσέγγισης. και από τις περιφερειακές αρχές. Στη Γαλλία, οι διοικητικές δομές είναι αρκετά περίπλοκες. Χρειάζεται κάποια απλοποίηση. Και σίγουρα η κυρία Ντελή και η κυρία Ροκόνη θα έχουν κάποιες συμπληρωματικές παρατηρήσεις για την επίσκεψη της αντιπροσωπείας μας στη Γαλλία. Πάντως, μας εντυπωσίασε η αποστολή αυτή. Ευχαριστώ. Η Σοφή Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ήταν μεγάλη τιμή μας να υποδεχθούμε την αντιπροσωπεία της Επιτροπής στη Γαλλία. Και θα μιλήσω για την δική μου περιοχή, την Τουρέν. Εκεί επισκεφθήκαμε με κάποιες επιχειρήσεις τεχνολογικές με υψηλή προσθέμενη αξία επιχειρήσεις που δεν παράγουν μαζικά, αλλά ασχολούνται με ειδικά τεχνικά προϊόντα, ιδιαίτερα στο σιδηροδρομικό τομέα. Πρόκειται για επιχειρήσεις που χάρη στα διαρθρωτικά ταμεία ξεπέρασαν και τις προσδοκίες τους για την καινοτομία και την τεχνολογική ανάπτυξη. Και στόχος ήταν να δείξουμε πώς οι περιφέρειες των κρατών μελών με υψηλό ΑΕΠ χρειάζονται ακόμη και σήμερα την οικονομική όθηση της περιφερειακής πολιτικής για να αναπτύξουν ε, οικονομική δραστηριότητα υψηλής προστιθέμενης αξίας και να δημιουργήσουν θέσεις απασχόλησης. Επίσης, ο τρόπος που αντιλαμβάνονται οι πολίτες τοπικά την περιφερειακή πολιτική δεν ανταποκρίνεται στην συμβολή της, στην πραγματική της συμβολή. Γιατί η περιφερειακή πολιτική είναι ευκαιρία της συγκεκριμενοποίησης, της ενσάρκωσης Ευρώπης στις περιφέρειες. Και έχουμε μία δημοσκόπηση του Ευρωβαρόμετρου που δείχνει πόσο απομακρυσμένοι αισθάνονται οι πολίτες από την Ευρωπαϊκή Ένωση και ιδιαίτερα στη Γαλλία η, περιφερειακή πολιτική μπορεί να γίνει ένας τρόπος στην Ευρώπη να συγκεκριμενοποιήσει τις δράσεις της στις συγκεκριμένες περιφέρειες επιτόπου. Και αυτό για τους τοπικούς παράγοντες και τους οικονομικούς φορείς. Η περιφερειακή πολιτική δεν έχει τη σωστή εικόνα που θα έπρεπε να έχει γιατί είναι δύσκολη στην εφαρμογή. Και μάλιστα ρώτησα έναν ιδιοκτήτη επιχείρησης αν είναι βαθμολογήσει από 0 στο 10, πόσο, πώς θα την περιπλοκότητα το, της πρόσβασης των προγραμμάτων, είπε 12. Φανταστείτε δηλαδή τι δρόμο έχουμε για να απλουστεύσουμε όλες αυτές τις διαδικασίες και τη γραφειοκρατία της περιφερειακής πολιτικής που κατά τη γνώμη μου είναι η πιο όμορφη ευρωπαϊκή πολιτική. Ευχαριστώ. Σον Κέλλη. Merci, euh, Madame la Κυρία Ντελή, συγγνώμη στην περιοχή Ile de France η αντιπροσωπεία ήταν πολύ αποτελεσματική. Αποτελεσματική γιατί είδαμε πώς είναι δυνατόν να έχουμε ολοκληρωμένα σχέδια με τη συμμετοχή πολλών παραγόντων και τοπικών φορέων και οργανώσεων και πολιτών. Και στο νησί Σεντενή με προγράμματα και σχέδια που καταδεικνύουν και την περιβαλλοντική και την κοινωνική διάσταση αλλά και το οικονομικό διακύβευμα. Σε τέτοιου είδου σχέδια είναι που αξιοποιήθηκε πραγματικά η περιφερειακή πολιτική. Σε ό,τι αφορά το urban, στο ΟΛΝΕ ναι, είδαμε ποια είναι τα απτά αποτελέσματα του προγράμματος Urban, που για την Ile de France δίνουν πραγματικά όθηση στην πολιτική των πόλων, με σφαιρική προσέγγιση, με συμμετοχική προσέγγιση, με ανάμειξη όλων των παραγόντων και με πολύ, αποτελεσμα... πολύ εντυπωσιακά αποτελέσματα. Στην περιοχή Λιντεφράν στη Γαλλία χρησιμοποιήθηκε το 4% του ΦΕΝΤΕΡ του Αναπτυξιακού Ταμείου με κονδύλια που στόχο έχουν ε, την ε, ανανέωση των πόλων με την ανακαίνιση των κτηρίων. Και μάλιστα ήταν ε, περίτρινη απόδειξη ότι όταν η πολιτική αξιοποιείται για να υλοποιήσει τις ε, ανάγκες και τα αιτήματα των πολιτών και να εισακούσει τις προσδοκίες του, τότε είναι που έχουμε μια πραγματική προστιθέμενη αξία της πολιτικής και θα πρέπει να συνεχίσουμε αυτή την πορεία. Τώρα έχει το λόγο ο Σον Κέλλη. Ευχαριστώ. Το μέλλον της χρηματοδότησης της συνοχής είναι ιδιαίτερα σημαντικό και στο παρελθόν και από εδώ και μπρος. Ένα ιδιαίτερα ενδιαφέρον σημείο είναι το ότι είναι σημαντικό και για τη μελλοντική χρηματοδότηση, αλλά και πιο σημαντικό το πώς θα περάσει αυτό το μήνυμα στους πολίτες. Η χειρότερη, ο χειρότερος μηχανισμός δημοσίων σχέσεων είναι η Ένωση σε όλο τον κόσμο. Γιατί οι πολίτες ακούνε μόνο τα κακά, ποτέ τα καλά. Η Σαμπίνα μας έδωσε ένα πολύ ωραίο παράδειγμα. Έγινε αξιολόγηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης από 0 έως 10, ως το πολύπλοκο, και έδωσε 12. Έτσι το αντιλαμβάνει ο κόσμος. Στη δική μου χώρα, τα τελευταία 15 χρόνια είχαμε μεγάλο μετασχηματισμό σε μεγάλο βαθμό λόγω κονδυλίων της Ένωσης και πιο συγκεκριμένα αυτής εδώ της Επιτροπή, δηλαδή περιφερειακά διορθωτικά κονδύλια. Το ξέρουν οι πολίτε, Όχι. Ήθελε ήθελη κυβέρνηση να το ξέρουν οι πολίτε, Όχι. Η κυβέρνηση ε, παρουσιάζεται το έκανε αυτή και η, η Ένωση δέχεται τα πειρά. Τώρα μπορεί να οδηγήσει κανείς από τον Μπέλφαστ στο βορρά μέχρι το Κόρκ στο νότο σε μεγάλο αυτοκινητόδρομο στην Ιρλανδία. Όταν άνοιξε αυτό ο δρόμο προημερών, ήταν παρουσία Ένωση. Όχι. Ξέρει ο κόσμο ότι η Ένωση έδωσε λεφτά. Όχι. Έχουμε μόνο μία πινακίδα που λέει εν μέρη χρηματοδοτήθηκε από την Ένωση. Μιλάμε λοιπόν για το μέλλον. Πρέπει επικοινωνιακά τα στοιχεία αυτά να δίνονται. Για το ίδιο το μέλλον της Ένωσης και τα δημοψηφίσματα κλπ. είδαμε ότι οι πολίτες έχουν αρνητική γνώμη για την Ένωση. Ενώ το μήνυμα θα έπρεπε να είναι θετικό. Γιατί έχουμε ξεδέψει και κονδύλια και χρόνο και έμφαση στις δημόσιες σχέσεις, αλλά δεν υποχρεώσαμε τι κυβερνήσει. Δεν το κάναμε αυτό. Όταν ένα πρόγραμμα χρηματοδοτείται από την Ένωση, η Ένωση να εκπροσωπείται όταν γίνεται τα εγγένεια, Και νομίζω εμείς ως Ευρωβουλευτές πρέπει να επιμένουμε σε αυτό. Το Ευρωκοινοβούλιο να εκπροσωπείτε σε οποιοδήποτε πρόγραμμα που χρηματοδοτείτε από την Ένωση. Και αυτό είναι δράση υπέρ της δημοκρατίας. Γιατί δείχνουμε στον κόσμο ότι η Ένωση λειτουργεί, αποδίδει, ενδιαφέρει για τους πολίτες και έχει ειδικό βάρος που μετράει. Αυτό δεν έγινε στο παρελθόν, πρέπει να γίνει από εδώ και μπρο. Ιωάχιμ Τσέλερα. Αγαπητοί συνάδελφοι, εδώ είναι σαν να καψουρίζουμε για τα δικά μας φάλματα. Μήπως να κοιτάξουμε λίγο και αυτά βεβαίως που έχουμε κάνει εμείς λάθος με στην ευρωπαϊκή πολιτική. Έχω και άλλα παραδείγματα θέλω να πω ότι δύο φορές πήγα στη Δυτική Πολωνία επισκέφθηκα σχολεία που από, αντίθετα από αυτά που μας λέτε εδώ, ε, ο κόσμος ήταν ενήμερος και μάλιστα ξέρανε και ποιος είναι ο βουλευτής της εκλογικής περιφέρειας. Ίσως αυτό έχει να κάνει βέβαια με την οργάνωση την εκλογική της Πολωνίας και τις εκλογικής περιφέρειες που υποχρεώνουν τον βουλευτή να είναι σε επαφή με τους ψηφοφόρους του, να μιλάει μαζί τους κτλ. Και βέβαια αντίστοιχα θα πρέπει να οργανώνουμε και τα χρονοδιαγράμματά μας, κοιτώντας όχι μόνο τι είδους εκδηλώσεις θα οργανώσουμε, αλλά και τι δουλειά μπορούμε να κάνουμε στην ουσία και στις εκλογικέ μας περιφέρειες ο καθένας. Θα ήθελα να ευχαριστήσω μεταξύ την κυρία, Ντελή, την κυρία και την κυρία Οκνίν για την επίσκεψη, γιατί ήμουν και εγώ μέλο τη αντιπροσωπεία στη Γαλλία. Έκαναν πολύ καλή δουλειά στην προετοιμασία τη επίσκεψη και έδειξαν ότι η συνοχή, η πολιτική τη συνοχή δεν, είναι, δεν κρίνεται μόνο από τι σχέσει πλούσιων και το ή δεν εκφράζει την αναλογία πλουσίων και φτωχών, αλλά πάνω απ' όλα το αποτελεί τον συνδετικό ιστό της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εδώ ακριβώς θα πρέπει να εντοπίσουμε τη δουλειά μας ε, στην ε, ανάγκη της αντιμετώπισης των προβλημάτων των μεγάλων αστικών κέντρων και των προαστιακών τους περιοχών με τις προτάσεις που έχουμε δει νομίζω ότι δίνονται καλές ιδέες και μια και πρόκειται να συστήσουμε την πολιτική συνοχής στο νέο γραφό στρατηγικής Ευρώπη 2020 Καταγράφεται βέβαια η πολιτική της συνοχής ε, ως ένα τομέα πολιτικής όμως ο οποίος ε, πρέπει πλέον να προχωρήσει από την απλή αναγνώριση κάποιων δεδομένων σε ουσιαστική πολιτική, σε πολιτική με περιεχόμενο γιατί αποτελεί κεντρική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Καλό θα ήταν να υπογραμμίσουμε ότι είχαμε μέχρι τώρα καλά αποτελέσματα ως προς την συνοχή, τη συνεκτική ανάπτυξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ότι εκεί που υπάρχουν ακόμη ανάγκες για δουλειά στη συνοχή πρέπει να βρούμε καινούργιες και καινοτόμους λύσεις και να μην περιοριστούμε μόνο σε αυτά που ήδη γνωρίζουμε. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Αν δεν θέλει κανένας άλλος να σχολιάσει θα μιλήσω κι εγώ ως μέλος της Επιτροπής. καλή ευκαιρία να καταλήξουμε και σε μερικά συμπεράσματα και να διδαχτούμε από τις μέχρι τώρα εμπειρίες. Ενθαρρύνω όλους τους συναδέλφους που θα οργανώσουν άλλα ταξίδια αλλού να διαβάζουν τις εκθέσεις για να παίρνουν ιδέες. Και κάτι άλλο. Όταν πάμε σαν βουλευτές σε μια περιοχή, σε μια πόλη, για να καταλάβουμε καλύτερα τα θετικά και τα αρνητικά της πολιτικής της Ένωσης για την οποία εξάλλου είμαστε συνυπεύθυνοι. Και η υποχρέωσή μας είναι αυτά τα ταξίδια να τα χρησιμοποιούμε για να αυξήσουμε την ορατότητα όπως υπόθηκε του Ευρωκοινοβουλίου. Είναι υποχρέασή μας με τη νέα συνθήκη. Και το Τμήμα Πληροφόρησης του Ευρωκοινοβουλίου θα μπορούσε να οργανώνει εκεί επί τόπου μια εκδήλωση για αυτό το στόχο. Θα μπορούσαν να το οργανώσουν την εκδήλωση αυτή όταν θα είμαστε εκεί και εμείς. Συμφωνήσαμε με τον Επίτροπο να υπάρχει πληροφόρηση όταν κάνει ένα ταξίδι να το συνδεύουμε και εμείς αν είναι στην εκλογική μας περιφέρεια. Το κάναμε στο παρελθόν αυτό. Βλέπω ότι ο Επίτροπος συμφωνεί. Οπότε μπορούμε να ζητάμε από το πολιτικό γραφείο του Επιτρόπου να μας το οργανώνει αυτό, κοινή αυτή η επίσκεψη στο μέλλον. Και με βάση απόφαση της διάσκεψης των Πρόεδρων θα στείλω την έκθεσή σας, έκθεσή σας στη διάσκεψη των Προέδρων των Επιτροπών. Να έχετε υπόψη ότι αυτές οι εκθέσεις δηλαδή θα τις διαβάσουν και άλλοι. Βάλτε λοιπόν μέσα όποια πληροφορία εσείς θεωρείτε χρήσιμη. Βανγίσταλ Ρόι. Δεν ήξερα ότι τόσοι πολλοί θα το διαβάζανε. Θα πρέπει να φροντίσουμε το έγγραφο να είναι ευανάγνωστο και πλήρες. Υπάρχει ένα άρθρο που με τα γελιά μου, ούτε και με τα γελιά μου δεν μπορώ να διαβάσω. Πρέπει να είναι βανάγνωστα. Πρόεδρος, ωραία. Ας προχωρήσουμε στο σημείο 6. Ένα σχέδιο γνωμοδότησης. Το έκανε η πρόεδρος. Σας θυμίζω τις αλλαγές στη νέα συνθήκη της νομοθετικής διαδικασίας. Έχω μια πρόταση της Κομισιόν για τους κανόνες και τις γενικές αρχές μηχανισμού ελέγχου από τα κράτη-μέλη της άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων της Επιτροπής. Μας ζητήθηκε γνωμοδότηση. Έχουμε αλλαγή στη συνθήκη ως προς το πλαίσιο των ε, εκτελεστικών αρμοδιοτήτων Νομοθέτης βέβαια είναι και το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο. Εμείς υποβάλαμε 16 τροπολογίες στο κείμενο Σάιερ της Νομικής Επιτροπής για το δικαίωμα πληροφόρησης του Κοινοβουλίου διαφάνεια επιλογή διαδικασιών και δικαίωμα του Κοινοβουλίου να αντιταχθεί στις εκτελεστικές αρμοδιότητες και άσκηση της εκ μέρους της Κομισιόν. Τεχνικονομικοί κανόνες, πολύπλοκοι. Υπάρχει προθεσμία κατάθεσης τροπολογιών 4 Ιουνίου. Πρέπει να ψηφίσουμε 21 με 22 Ιουνίου. Η νομική ψηφίζει στις 23 Ιουνίου. Αυτή είναι η μόνη απόφαση που πρέπει να πάρουμε. Η γραμματεία μπορεί να σα βοηθήσει με τι τροπολογίες. Σχόλια. Περνάμε στο σημείο 7. για ένα θέμα που ήδη έχουμε πάρει απόφαση, αλλά με τη νέα συνθήκη το Συμβούλιο εισήγαγε αλλαγέ. οπότε χρειάζεται νέα διαδικασία διαβούλευσης με το Ευρωκοινοβούλιο Συναντήσαμε την νομική υπηρεσία του Συμβουλίου Ζητήσαμε και τη γνώμη δικό, της δικής μας νομικής υπηρεσίας. Όλα αυτά με την απλουστευμένη διαδικασία όπως χρησιμοποιούσαμε, τη χρησιμοποιούσαμε πριν, δηλαδή χωρίς τροπολογίες. θα κλείσουμε με το θέμα αυτό μέσα στον Ιούνιο. Χρειάζεται σύσταση των συντονιστών. Η πρόεδρος ορίστηκε ως εισηγήτρια. Για την επαναδιαβούλευση μπορούμε να διαλέξουμε. Είτε παραμένει η πρόεδρος, η εισηγήτρια ή τη βάζουμε άλλον. Αυτή είναι η μόνη απόφαση. Σχόλια. Ωραία, θα το ρυθμίσουν, θα κάνουν τη σύσταση συντονιστές. Ελπίζω να ήρθε ο κύριος Ντίρκ Άνερ. Μπορούμε να αρχίσουμε πέντε λεφτά πιο νωρίς. Με το σημείο 8. Είναι ο Γενικός Διευθυντής για την Περιφερειακή Πολιτική. Επίσης η Βερόνικα Γκάφη. Τη γνωρίσαμε στην πρώτη φάση αξιολόγηση 2000-2006. Τώρα είναι επικεφαλής προϊσταμένη του τμήματος αξιολόγησης. Ελάτε εδώ στο Προεδρείο. Um, uh, dear colleagues, uh, you might remember that when we had the, the previous exchange of views. Θα θυμόσαστε συνάδελφοι όταν συζητήσαμε το θέμα αυτό με την κυρία Γκάφη και την κυρία Κατερίνα Ματέρνοβα, κάπου εκεί Σεπτέμβριο-Οκτώβριο, είμαστε στην πρώτη φάση της έκθεσης αξιολόγησης. που έχει ξεκινήσει η Γενική Διεύθυνση Ρέτζι 2000-2006. Κυρίως για το, για το Περιφερειακό Ταμείο Οπότε ε, αναφερθείτε όλες και σε άλλου είδου χρηματοδότηση. Η εξολόγηση έχει ολοκληρωθεί. Είναι σημαντική για μας για τις μελλοντικέ υποθέσεις. Βέβαια και η Κομισιόν και το Κοινοβούλιο υποφέρουμε, γιατί εξολογούμε το 2006 για να βγάλουμε πορίσματα 2014-2020. Τι να κάνουμε. Αφού δεν έχουμε άλλα στοιχεία από την τρέχουσα περίοδο. Παρακαλώ τον Dirk Άνερ να πάρει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Καλησπέρα σε όλα τα μέλη της Επιτροπής Περιφερειακής Πολιτικής. Θα ήθελα καταρχάς κυρίες και κύριοι να σας ευχαριστήσω θερμά που μας δίνετε σήμερα αυτή την ευκαιρία να παρουσιάσουμε τα αποτελέσματά μας για την περίοδο 2000-2006 ως προς το Περιφερειακό Ταμείο. Θα έχουμε, πιστεύω, σε μερικούς μήνες αντίστοιχα την επισκόπηση για το Ταμείο Συνοχής και αργότερα και το, ταμείο, το Κοινωνικό Ταμείο. Βλέπουμε λοιπόν αυτή την αξιολόγηση ως μια πολύ σημαντική συνεισφορά σε έναν διάλογο ελεύθερο σε ένα, με ένα, μαζί με ένα ευρύτατο κοινό και γι' αυτό χαίρομαι ιδιαίτερος για την ευκαιρία που μας δίνεται να σας παρουσιάσουμε σήμερα τα αποτελέσματα αυτής της μελέτης, γιατί είστε οι κύριοι εταίροι μας ως προς το, η χάραξη πολιτικής και την παρακολούθηση της εφαρμογής αυτής. Ποτέ μέχρι τώρα πρέπει να πω δεν είχε επενδυθεί τόσο πολύ σε μια εκ των εξτέρων αξιολόγηση όπως τώρα για την περίοδο 2000-2006 επενδύσαμε τόσο πολύ γιατί θέλαμε τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα. Ήμασταν σε γνώση δηλαδή ότι αυτή θα ήταν η μόνη μα αξιολόγηση πάνω στην οποία θα μπορούσαμε να στηριχθούμε, από την οποία θα μπορούσαμε να διδαχθούμε για την περίοδο μετά το 2013. Και έτσι αλλάζουμε σε σχέση με τις προηγούμενες αξιολογήσεις την προσέγγιση μας. Στο παρελθόν προσπαθούσαμε να κάνουμε την εκ των αξιολόγηση με μια ολιστική μάλλον προσέγγιση με μια μεγάλη δηλαδή μελέτη ε, αξιολόγηση προσπαθούμε να καταγράψουμε κάθε είδους αντίκτυπο και αποτελέσματα των πολιτικών μας. Τα αποτελέσματα αυτά, μάλλον η προσέγγιση αυτή, απεδείχθη μη ικανοποιητική. Ήταν υπερβολικά ευρεία. Τα δε αποτελέσματα ήταν ασαφή και γενικά. Σε υπερβολικό βαθμό. Τώρα λοιπόν προτιμήσαμε να επιλέξουμε μια διαφορετική προσέγγιση ε, διτά διαφορετική. Πρώτον, διότι χωρίζουμε τη συνολική περίοδο σε θεματικές ενότητες, στις οποίες θα αναφερθώ ευθύς αμέσως, και δεύτερον, διότι για κάθε ένα από τα θέματα, από τους τομείς πολιτικής, της περιφερειακής πολιτικής, ορίσαμε, συγκροτήσαμε μια ομάδα εμπειρογνωμόνων, η οποία ανέλαβε την αξιολόγηση έτσι ώστε από κοινού με αυτούς να προσδιορίσουμε τη βέλτιστη δυνατή μέθοδο αξιολόγησης για τον συγκεκριμένο τομέα. Αυτό βέβαια εξαρτώνταν πάντα από τις πληροφορίες και τα δεδομένα που είχαμε στη θέση μας, αλλά και από το αντικείμενο μελέτης, το συγκεκριμένο τομέα δηλαδή. Ο κύριος μας στόχος εκ τούτου ήταν να έχουμε όσο το δυνατόν πιο συστηματικά σωστές πληροφορίες για τους κύριους τομείς πολιτικής. Με ένα απλό σκεπτικό, δηλαδή να έχουμε τον καλύτερο εμπειρογνώμονα, την καλύτερη τεχνογνωσία, τις καλύτερες μεθόδους και ως εκ τούτου αναπτύχθηκε μέγα φάσμα διαφορετικών μεθόδων και δειγματοληπτικές μελέτες και μακροοικονομικά πρότυπα και δειγματοληπτικές ε, ε, ή υποθέσεις ε, σε πραγματικά περιστατικά και έτσι προσπαθήσαμε βάσει αυτών να ε, μελετήσουμε ένα πρακτικό θέμα εντό εισαγωγικών περιφερειακής πολιτικής. Γιατί βεβαίως θα πρέπει δυστυχώς να επισημάνω ότι δεν υπάρχει ένας μόνο δείκτης που να επαρκεί για να παρατηρηθεί αν ήταν ή όχι επιτυχής η πολιτική συνοχής τα θέματα για την αξιολόγηση, τα ερωτήματα μάλλον για την αξιολόγηση ήταν πολύ συγκεκριμένα. Τι συγκεκριμένα έχει γίνει έτσι ώστε να καλυφθούν οι διαφορέ στην ανάπτυξη, τι έχει επιτευχθεί σε συγκεκριμένου τομεί πολιτική και θα δείτε από τι διαφάνειε που σα έχουμε μοιράσει τι διάφορε απαντήσει, το input. Έχουμε αυτό που ονομάζουμε modeling block, εκεί δηλαδή που χρησιμοποιούμε διάφορα μακροοικονομικά μοντέλα για να δούμε σε ποιο βαθμό η ανάπτυξη που παρατηρείται σε συγκεκριμένες περιοχές σύγκλησης κατά την χρονική αυτή περίοδο μπορεί να ερμηνευθεί, να αποδοθεί στην πολιτική συνοχής. Πέραν αυτού όμως του συστήματος, της προσέγγισης με τα μοντέλα, έχουμε και άλλα συστήματα εφαρμογής τα οποία μας δίνουν πολύτιμες πληροφορίες. πριν ξεκινήσουμε τη μεγάλη αυτή αξιολόγηση, είχαμε ορίσει μεγάλες ομάδες ε, δικτών, συντελεστών, που θα μπορούσαν να καταγραφτούν, να αξιοποιηθούν μάλλον, για να ε, εκτιμήσουμε διαφορετικά project. Όλα αυτά προσπαθήσαμε να τα καταγράψουμε για την πρώτη προσέγγιση, για το ΦΕΟΓΑ και με βάση τις θεματικές ομάδες που είχαμε επιλέξει, που τις βλέπετε στο κάτω μέρος αυτής της ε, διαφάνειας, της σελίδα που είναι υποστήριξη επιχειρήσει στο περιβάλλον και κλιματική αλλαγή, το, οι μεταφορές, διαφορετικέ αλλαγές και η παγκοσμιοποίηση, ε, ισότητα μεταξύ των φύλων, η εκπροσώπηση των φύλων και δημογραφικά στοιχεία, περιφερειακή ανάπτυξη. Όπως βλέπετε, είχαμε τις πρωτοβουλίες, ε, τις κοινωτικές πρωτοβουλίες Interreg και Urban, και θα έχουμε σύντομα και για το Ταμείο Συνοχής τα τελευταία στοιχεία, το οποίο το Ταμείο Συνοχής καθυστέρησε. Γιατί βέβαια, καθέσει η εξολόγησή του, γιατί άρχισε πιο αργά η εφαρμογή του και διαρκεί και περισσότερο. Γι' αυτό προσπαθούμε να έχουμε στο δυνατόν, προσπαθώντας να έχουμε περισσότερες πληροφορίες, ε, καθυστερήσαμε την ε, διαδικασία της αξιολόγησης του Ταμείου Συνοχής. Εάν μου επιτρέπετε τώρα, θα ήθελα να παρακαλέσω τη συνάδελφο Βρόνικα Γκάφη, που είναι επικεφαλής της ομάδας αξιολόγησης, να μας καθοδηγήσει στην ανάγνωση των αποτελεσμάτων αυτής της μεγάλης... Α, εσείς όμως δεν θα φύγετε, λέει η κυρία Χιούμπνερ. Όχι, όχι, λέει ο κύριος Άνερ, με χαρά θα μείνω κοντά σας. Η κυρία Γκάφη, ευχαριστώ πολύ Ντέρκ, ευχαριστώ κυρία Χιούμπνερ που με προσκαλέσατε και εμένα εδώ σε αυτή τη συνεδρίαση της Επιτροπής Περιφερειακής Πολιτικής να σας παρουσιάσω τα αποτελέσματα της αξιολόγησής μας. Όπως σας είχαμε υποσχεθεί, ξαναρχόμαστε για να σας δώσουμε τα πλήρη αποτελέσματα της ε, αξιολόγησης. Θα προσπαθήσω να σας δώσω τα κύρια πορίσματα από την ε, συνθετική έκθεση, η οποία πρέπει να επισημάνω συνοψίζει το έργο των 14 ομάδων αξιολόγησης των εμπειρογνωμόνων και τρία χρόνια δουλειάς. 4,2 εκατομμύρια ευρώ κόστησε η αξιολόγηση. Μήνυμα λοιπόν που απορρέει από όλα αυτά είναι ότι ναι, κοστίζει γιατί την αξιολόγηση μπορεί να μην δίνονται απαντήσει σε όλα τα ερωτήματα μεν, αλλά τέτοιου είδους προσπάθεια και στήριξη χρειάζεται για να έχουμε συγκεκριμένα αποτελέσματα των προσπαθειών μας. Έχουμε την έκθεση στην διάθεσή σας, στην ε, είσοδο της αίθουσας. Εάν τυχόν δεν φτάνουν τα αντίτυπα, πολύ ευχαριστώ να σας κάνουμε φωτοτυπίες ή να σας διαθέσουμε περισσότερα αντίγραφα αν χρειάζεται. Για να δούμε λοιπόν τι έγινε στην περίοδο 2000-2006. Για να περάσουμε μετά στο ερώτημα σε τι συνεισέφερε, σε ποιο βαθμό συνεισέφερε η περιφερειακή η πολιτική συνοχή. 2000-2006 λοιπόν σημειώνεται υψηλότερη ανάπτυξη στην, ε, στις περιφέρειες του στόχου 1. Στην, ε, στους 25 της Ευρωπαϊκής Ένωσης μειώνονται περιφερειακές αποκλήσεις, στους 15 της Ευρωπαϊκής Ένωσης πλην της Ελλάδας και αυτό έχει να κάνει με την ανάπτυξη της περιοχής της Ελλάδας, της περιοχής Αθήνας, συγγνώμη, ε, μειώνονται οι αποκλήσεις. Στην Ευρώπη των 10 ευρύνονται, διευρύνονται οι αποκλήσεις λόγω υψηλής ανάπτυξης της ε, ε, πρωτεύουσα και στο στόχο 1 στην Ευρώπη των 15 είχαμε 2% ανάπτυξη στο ΑΕΠ κατά κεφαλή, 1,4% στις περιφέρειες που δεν είχαν την αντίστοιχη στήριξη. Βλέπουμε δηλαδή γενικά θετική εξέλιξη στην Ευρώπη, χωρίς όμως να μας δίνει αυτό επαρκή εικόνα του σε τι βαθμό συνεισέφερε η πολιτική συνοχή στην ανάπτυξη αυτή. Και όπως λέμε σε αυτήν εδώ την ε, διαφάνεια, δεν μπορούμε την επιτυχία, την, ε, τον βαθμό επιτυχίας της πολιτικής αυτής να τον ε, αξιολογήσουμε μόνο με την παρατήρηση των στατιστικών στοιχείων. Άρα χρειάζεται να δούμε και άλλα ζητήματα, άλλα ερωτήματα, εάν ήταν επαρκής η κλίμακα της χρηματοδότησης, εάν ήταν στοιχευμένη σωστά στους κατάλληλους παράγοντες, εάν τα μακροοικονομικά μοντέλα δίνουν ε, επαρκείς ενδείξεις ανάπτυξης. Εάν οι επιδιώσεις στην ανάπτυξη ήταν καλύτερες στις περιοχές που στηρίχθηκαν από την πολιτική συνοχή και αν υπάρχουν συγκεκριμένα στοιχεία, αποδείξεις δηλαδή θετικών αποτελεσμάτων. Σε όλα αυτά τα ερωτήματα ευτυχώς η διαπάντηση είναι θετική. Είχαμε δηλαδή σημαντική βελτίωση στις ε, περιοχές του στήριξης, ιδιαίτερα στο στόχο 1 με 2-3%, 2 με 3% συνολικών προσδορισμένων επενδύσεων στις περιφέρειες του στόχου 1 και με την ε, ιδιωτική επένδυση, 1% του επανάπτυξη στην Ελλάδα και την Πορτογαλία. Επίσης γνωρίζουμε από τις αξιολογήσεις ότι το ΦΕΟΓΑ στόχευε ιδιαίτερα τους παράγοντες ε, ανάπτυξης που έχουν εντοπίσει όλες συνολικά οι πολιτικές, οι πολιτικές οικονομίες, δηλαδή συνοχή και υποδομές. Εάν κοιτάξουμε λοιπόν λίγο την κλίμακα, τις επενδύσεις και τις υποδομές, εάν κοιτάξουμε την ε, κλίμακα, ε, στις ε, δαπάνες της πολιτικής συνοχής σε σχέση με, τη συνολική, με τους συνολικούς μέσους όρους αναέτος των, επί του ΑΕΠ, βλέπουμε ότι στην Ευρώπη των 15 είναι 7,28%, στην Ευρώπη των 10 είναι 14,37%, δηλαδή σημαντικό ποσοστό επί, του ΑΕΠ εκπροσωπούν οι πόροι της συνοχής. Και προχωρούμε με το πρότυπο, με μοντέλο Quest, για να μην έχουμε πολλούς παράγοντες και μπερδευτεί η περισσότερη εικόνα. Κοιτούμε συνολικά την ε, ανταπόκριση επί του ΑΕΠ. Στην Ευρώπη των 25 για την περίοδο 2000 με 2009 έχουμε σορευτικό καθαρό αποτέλεσμα επί του ΑΕΠ της πολιτικής συνοχής σε επίπεδο 0,7% το οποίο για το 2000 με 2015 ανέρχεται σε 2,4% και αντίστοιχα υψηλά ποσοστά βλέπουμε στην Ευρώπη των 10, 3,7, 10,2 και κάπως χαμηλότερα για την Ευρώπη των 15, 0,5, 1,9. Πάντως αυτό στηρίζεται στο μοντέλο, γιατί το μοντέλο στηρίζεται στις θεωρίες για τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί η οικονομία και πάνω σε αυτά τα δεδομένα προχωρούμε στην ανάπτυξη των μοντέλων μας, ε, με, με, δεδομένο ότι εκεί πέρα πρέπει να συμβάλλει η πολιτική συνοχή. Πρέπει να επισημάνω όμως ότι υπάρχει και ένα άλλο μοντέλο, το μοντέλο Herman, το οποίο έχει διαφορετική διάρθρωση, κατασκευή, δεν συμφωνούν πάντοτε τα μοντέλα μεταξύ τους, αλλά και τα δύο μοντέλα που είδαμε μας αποδεικνύουν, μας πείθουν ότι έχει θετική, θετικό αντίκτυπο επί του ΑΕΠ η πολιτική συνοχή. Στην προ, επόμενη διαφάνεια βλέπετε την διάρθρωση των επενδύσεων, μόνο και μόνο για να σας επισημάνουμε ότι διαφορετικές στρατηγικές φέρνουν διαφορετικά αποτελέσματα σε κάθε περιοχή της Ευρώπης. Το πράσινο είναι εκεί που έχουμε περισσότερες επενδύσεις στις βασικές υποδομές. Το πράσινο δείχνει τις περιοχές που έχουν περισσότερη παραγωγή, περισσότερο παραγωγή περιβαλλοντική. Το κόκκινο είναι ανθρώπινη πόροι και το άλλο χρώμα έχει μεγαλύτερο μείγμα ε, επενδυτικό. Άρα βλέπουμε διαφορετικές στάσεις ως προς τις επενδύσεις σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση και βέβαια αυτό έχει να κάνει και με το ΦΕΟΓΚΑ και με το Ταμείο Συνοχή. Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο δεν συμπεριλαμβάνεται στην διαφάνεια που βλέπετε εδώ. Και βλέπετε ω εκ τούτου με, ε, με γραφική αναπαράσταση πώ επενδύονται οι πόροι. Για να περάσω τώρα στι θεματικέ ενότητε, πρώτα απ' όλα περνάω στην στήριξη των επιχειρήσεων όπου τα κράτη-μέλη καταγράφουν δημιουργία πάνω από ενό εκατομμυρίου θέσεων εργασία χάρη στη στήριξη τη επιχειρήση. Πολύ μεγάλα ποσοστά, πιθανόν να έχουν όντω επιτευχθεί, αλλά δεν είναι πλήρη και δεν είναι απολύτω ακριβή. Γιατί, διότι ορισμένα κράτη-μέλη μας δίνουν πολύ καλά συστήματα, έχουν πολύ καλά συστήματα καταγραφής και αποδόση δεδομένων, με ουσιαστική καταγραφή των δεδομένων και επισημαίνω εδώ ιδιαίτερο στη Ηνωμένο Βασίλειο και τη Γερμανία ως καλά παραδείγματα, ενώ υπάρχουν κάποια άλλα τα οποία δεν καταβάλουν το ίδιο, καλές, ε, το ίδιο έντονες προσπάθειες για να καταγράψουν τη δημιουργία θεσμών εργασία ε, χάρη στην ε, στήριξη των επιχειρήσεων. Άρα μπορεί κάπου να καταγράφονται υπερβολικά πολλέ θέσει εργασία και σε κάποια άλλα σημεία να μην είναι επαρκή η καταγραφή. Πάντω, συνολικά η εικόνα που μα δίνεται από όλα μα τα προγράμματα στην στήριξη των επιχειρήσεων είναι αρκετά κοντά σε αυτήν που βλέπετε εδώ. Προσπαθούμε επίση να καταγράψουμε τι νέε μεθόδου αξιολόγηση και να χρησιμοποιήσουμε τι καλύτερε ε, ε, μεθόδου αξιολόγηση των επενδύσεων ανεργαζόμενο και ιδιαίτερα να, να εκτιμήσουμε την, ε, τις επιδόσεις μιας υποστηριζόμενης επιχείρησης σε σχέση με αυτές ε, τις επιχείρηση, η οποία δεν έχει τέτοια στήριξη. Βέβαια εκ των υστέρων είναι πιο δύσκολο να γίνει η αξιολόγηση, ειδικά αν δεν έχει προγραμματιστεί εξάντε και όταν δεν υπάρχουν επαρκή δεδομένα. Παρόλα αυτά όμως έχουμε για την Ανατολική Γερμανία υψηλότερε επενδύσεις ανεργαζόμενων στις επιχειρήσεις που είχαν τη στήριξη συγκρινόμενες με εκείνες που δεν είχαν στήριξη. 11, με 11 ευρώ 11 με 12.000 ευρώ επενδύσεις αντί για 4.000 ευρώ. Και μάλιστα από μια συνεδρία σήμερα το πρωί με εμπειρογνώμονε από την Ιταλία, τη Σουηδία και το Ηνωμένο Βασίλειο, με του οποίου είχαμε μια ανταλλαγή απόψεων για τι ιδέε που θα μπορούσαμε να αναπτύξουμε για το μέλλον, γιατί εδώ ακριβώ βλέπουμε ότι χρειάζεται περισσότερη προσπάθεια και θα θέλαμε και από τα κράτη-μέλη αντίστοιχα να δούμε περισσότερη προσπάθεια. Βλέπουμε πω η μέθοδο αξιοποιεί οικονομετρικέ μεθόδου βέβαια μας δίνει και πιο ικανοποιητικά αποτελέσματα και θέτει και ζητήματα πολιτικής. Η υποστήριξη λοιπόν των επιχειρήσεων ως αποτέλεσμα αυτής της αξιολόγησης και στην τελική φάση ζητούμε, ρωτούμε είναι προ συζήτηση φυσικά όλο αυτό, πρέπει να συζητήσουμε, πρέπει να συζητήσουμε τα κράτη-μέλη. Εάν θα πρέπει να δίδεται στήριξη στι μεγαλύτερε επιχειρήσει ή αν αρκεί να δραστηριοποιηθούν μόνε του και να κάνουν σχετικέ επενδύσει μόνε στι μεγάλε επιχειρήσει. Βέβαια, για να δοθεί τελική απάντηση, πιστεύω, θα πρέπει να έχουμε περισσότερε προσπάθειε ώστε την αποτελεσματικότητα διαφόρων μορφών στήριξη στι επιχειρήσει. Αυτό μπορούμε να το κάνουμε ε, όλοι μαζί, δεν είναι κάτι που μπορούμε να κάνουμε μόνο μας επί Ευρωπαϊκής Επιτροπής, πρέπει μαζί με τις περιφέρειες να κάνουμε πιο αυστηρούς, με πιο αυστηρούς κανόνες και μεθόδους αξιολόγηση των διαφόρων επενδύσεων και παρεμβάσεων προ επιχειρήσεις. Το τέταρτο ερώτημα έχει να κάνει με τις, πιο, με τις ορθές μεθόδους στήριξη και μάλιστα κατά την προετοιμασία αυτή τη παρουσίαση μέχρι το βράδυ, είχα ξαφνικά την ιδέα ότι σωστά ήταν καλό να ε, καταγράφουμε και την διαφύλαξη θέσεων εργασία, γιατί μιλούμε εδώ και χρόνια για τη διαφύλαξη θέσεων εργασία, αλλά δεν είναι αυτό μέτρο υπολογισμού τη αποτελεσματικότητα μια πολιτική. Μπορεί στη δεκαετία του 90 να είχαμε την προσπάθεια να διαφυλάξουμε θέσει εργασία, ενώ τώρα, στον 21ο αιώνα, στρεφόμαστε μάλλον προ τη δημιουργία νέων θέσεων εργασία και θέσεων εργασία σε νέου τομεί στην, ε, στους χώρους της οικονομίας που έχουν υψηλή ένταση γνώσης. Ε, και βέβαια είναι πολύ δύσκολο μερικέ φορέ να γνωρίζει κανεί τι σημαίνει διαφύλαξη εργασία ε, και αν είναι σκόπιμο το, ότι όντι με στήριξη να ε, συμβάλλουμε στην διαφύλαξη τη εργασία. Νέε λοιπόν θέσει εργασία, αυτέ που προσπαθούμε να καταγράψουμε και να υπολογίσουμε. Ε, πρέπει να συζητήσουμε όμως πώς, πότε, υπολογίζονται οι νέε θέσει εργασία και καταγράφονται οι νέε θέσει εργασία που δημιουργήθηκαν, γιατί υπάρχει μια διαφορά μεταξύ των δημιουργηθισών νέων θέσεων και τη ενίσχυση τη παραγωγικότητα. Φυσικά αυτό πάλι έχει σημασία να το δούμε για να δούμε τι είδου ε, στήριξη προσφέρουμε. Δηλαδή, το να λέμε ότι κάνουμε επένδυση σε μια επιχείρηση, δημιουργούνται νέε θέσει εργασία για εκείνου που θα κληθούν φερρυπίν να χειριστούν τον νέο εξοπλισμό τον οποίο αφορά η επένδυση και μακροπρόθεσμα έχουμε περισσότερη ε, παραγωγικότητα. Όμω αυτό μπορεί να έχει και αντίστροφο αποτέλεσμα. Δηλαδή μπορεί να γίνει επένδυση σε εξοπλισμό, η οποία επένδυση να έχει σαν αποτέλεσμα να μην χρειάζονται αρκετέ θέσει εργασία πλέον στην επιχείρηση, που ταυτόχρονα όμω μπορεί να οδηγήσουν μακροπρόθεσμα σε επέκταση του κύκλου εργασιών και άρα σε ανάγκη για περισσότερε θέσει εργασία. Δεν υπάρχει επομένω μία λύση η οποία να, είναι, ε, να, να ταιριάζει σε όλα τα νούμερα μεταφορές. Και πώς συμβάλλει το ΦΕΟΓΑ στις μεταφορές, το οποίο χρηματοδοτεί το 13%. Το ΦΕΝΤΕΡ το 13% όλων των ε, ε γραμμών υψηλή ταχύτητα, 24% τη επέκταση των αυτοκινητοδρόμων. Και άρα χρηματοδοτεί 26% των 7.734 χιλιόμετρων αυτοκινητοδρόμων που ολοκληρώθηκαν στην Ευρώπη των 15 και την αναβάθμιση των 3 χιλιόμετρων των σιδηροδρομικών γραμμών αντίστοιχα. Δοκιμάσαμε λοιπόν το μοντέλο. Προσπαθήσαμε να χρησιμοποιήσουμε το μοντέλο TransTools από το Κοινό Κέντρο έρευνα τη Σεβίλη, Σεβίλης, ε, το οποίο όμω δεν μας έδωσε τα αναμενόμενα αποτελέσματα, γιατί θέλαμε να δούμε και τα επιπτώσει επί του ΑΕΠ, αλλά και επί του περιβάλλοντος. Θέλαμε λοιπόν ένα νέο μοντέλο, με δεδομένα ίσως του Ταμείου Συνοχής να είναι πιο ξεκάθαρη η εικόνα, όταν τα έχουμε έτοιμα. Πάντως, το Transtools απαιτεί να έχει κανεί συνολικά έναν αυτοκινητόδρομο ολόκληρο από το ένα σημείο στο άλλο ή μια σιδηροδρομική γραμμή από το ένα σημείο στο άλλο και όχι διάφορα τεμάχια τμήματα αυτοκινητόδρομου ή σιδηροδρομικού. Φυσικά υπάρχουν ζητήματα που ακόμη πρέπει να επιληθούν, ενδεχομένω να πρέπει να μελετηθούν περισσότερο, να ληφθεί η δράση. Οι σιδηροδρομικέ γραμμέ υψηλή ταχύτητα, σε παραδείγματι, που είχαν γεννήσει αρκετά ζητήματα και ερωτηματικά και δεδομένου του υψηλού του κόστου και αμφισβητούμενε ε, αμφισβητούμενο αντίκτυπο στις ε, περιφέρειες. Ε, ζητήματα επίσης είχαν τεθεί ως προς τους λιμένες και τους αερολιμένες. Η σύσταση έλεγε να κοιτάξουμε περισσότερο την πρόσβαση στους λιμένες και τους αερολιμένες και να μην προσπαθήσουμε να ε, χρηματοδοτήσουμε πράγματα τα οποία καλύπτει ούτως ή άλλως από μόνη της η αγορά και Βέβαια πρέπει να πω ότι προχώρησαμε περισσότερο από τη αξιολόγηση εδώ, γιατί φτάνουμε να διατυπώσουμε ένα ερώτημα για το αν θα πρέπει στην Ευρώπη των 15 πλέον να χρηματοδοτείται η κατασκευή δρόμων. Στην Ευρώπη των 12 είναι ξεκάθαρο ότι χρειάζεται αναβάθμιση, προσπάθεια για την αναβάθμιση των οδικών αρτηριών, για τη βελτίωση οικονομική ζωή, για τη βελτίωση των συνδικών ασφαλεία κτλ. Αλλά το κατά πόσον χρειάζεται να κατασκευαστούν νέοι δρόμοι και με δεδομένη την τάση για περισσότερο πράσινες επενδύσεις, για περισσότερες πράσινες επενδύσεις, είναι αμφιδισβητούμενο το αν θα πρέπει να σχεδιαστούν και να κατασκευαστούν περισσότεροι δρόμοι. Τώρα, ε, η κοινωνική και εδαφική συνοχή, για να περάσω στο επόμενο κεφάλαιο, ε, διότι με την μελέτη αυτή είδαμε το εξή ότι μερικές φορές τα βάζουμε όλα μέσα σε ένα ε, πακέτο και θεωρούμε ότι πάντοτε τα πάντα αφορούν την κοινωνική συνοχή. Όχι, δεν είναι τα πάντα κοινωνική συνοχή, ε, είναι και οικονομική συνοχή και κοινωνική και εδαφική συνοχή. Και πράγματα τα οποία ενδεχομένω να μην προσφέρουν οικονομική ανάπτυξη έχουν μεγάλη σημασία για την κοινωνική και την εδαφική συνοχή. Και άρα πρέπει και αυτά να καταγραφούν. Ένα τρίτο λοιπόν του στόχου 1 του ΦΕΝΤΕΡ και 36% του στόχου 2 είχε να κάνει με τις κοινωνικούς στόχους και την εδαφική την εξορρόπηση των εδαφικών διαφορών, μάλλον και όχι την οικονομική ανάπτυξη. Άρα δεν μπορούμε να λέμε ότι αν δεν, υπάρχουν, αν δεν υπάρξει μείωση των ε, οικονομικών διαφορών έχει αποτύχει το σχέδιο, έχει αποτύχει η χρηματοδότηση, διότι μπορεί να έχουμε καλά αποτελέσματα στη συνοχή, την κοινωνική και την εδαφική. Κύρια λοιπόν ε, μετρήσιμα στοιχεία ήταν οι υποδομές, ο σχεδιασμός και η αποκατάσταση, ανάπτυξη δηλαδή ε, συνθήκων παροχής ε, καθαρού πόσιμου νερού για 14 εκατομμύρια κατοίκους επιπλέον, σε νοικοκυριά δηλαδή των ε, μειονεκτικών περιοχών, ή αποχέτευσης για πάνω από 20 εκατομμύρια κατοίκων, ανακαίνιση, αναζωγόνηση χωριών, κέντρων μεγάλων του κέντρου μεγαλοναστικών κέντρων, παλαιών βιομηχανικών εγκαταστάσεων ή ε, χώρων εθνικής πολιτιστικής κληρονομιάς. Και για να σας δώσω μια ιδέα, από τη σημερινή μας συνεδρία στο πρωί, μας δώσαν ένα παράδειγμα. Βορειοανατολική Αγγλία. Μία γερμανική ε, εταιρεία πήγε να εγκατασταθεί στην Ανατολική Αγγλία και ζητήθηκε να δώσει στοιχεία για το πόσε θέσει εργασία θα δημιουργούσε επιπλέον. Ρωτήθηκε γιατί επέλεξε την περιοχή αυτή κτλ. Και η απάντηση που έδωσε ήταν πάνω απ' όλα η ανακαίνιση η δυνατότητα της αναζωογόνησης της πόλης, η βελτίωση της ποιότητας ζωής, όπως τα λέγαμε συνοπτικά. Που βέβαια μπορεί να μην έχει άμεσα οικονομικά αποτελέσματα, αλλά πάντως σημαντικά. Βλέπουμε λοιπόν και παρατηρούμε όταν μελετούμε τις διάφορες περιπτώσεις και αποστέλουμε τα έντυπα για την αξιολόγηση όλη την Ευρώπη και βελτίωση στην ε, ποιότητα ζωή και τι εδαφικέ ισορροπίε ή κάλυψη των ανισοτήτων, χωρίς όμως να έχουμε συγκεκριμένα στοιχεία επαρκή για να κάνουμε μετρήσει. Πρέπει να μελετήσουμε περισσότερο αυτή την υπόθεση και πάλι ίσω ένα δείκτης να μην αρκεί. Δηλαδή να βρίσκαμε ένα δίκτυο ο οποίο θα αρκούσε να μπει στο σύστημα τη Eurostat για να μα δώσει αποτελέσματα συγκεκριμένα. Ίσως είναι αυτό ακόμα. Βλέπουμε σημαντική βλέπουμε περιορισμένη μάλλον, περιορισμένο αντίκτυπο προς την ανάπτυξη, αλλά ενισχυμένες συνθήκες αηφόρου ανάπτυξης και μείωση των κοινωνικών και εδαφικών διαφορών συμπεράσματο προ την πολιτική ότι τα επιτεύγματα τη πολιτική συνοχή ξεπερνούν μόνο την απλή και μόνο οικονομική ανάπτυξη, δηλαδή πρέπει να μιλούμε για πολλαπλού στόχου και επίση θα πρέπει να ξεκαθαρίσουμε τι θέλουμε να επιτύχουμε τη χρηματοδότηση του ΦΕΝΤΕΡ και ποιο είναι, ποιος είναι ο σύνδεσμο, ποιο είναι ο σχετισμό με την περιφερειακή ανάπτυξη. Όταν δηλαδή αποφασίζεται να γίνει επένδυση σε τέτοιου είδου περιοχέ παρέμβαση. Ε, καλό θα είναι να έχουμε σαφή εικόνα και να ακολουθούμε μια ξεκάθαρη λογική του τι κάνουμε και γιατί, τι θέλουμε να αλλάξει δηλαδή σε μια συγκεκριμένη περιοχή. Αν δούμε ιδιαίτερα το, την περίπτωση του στόχου 2, ε, όπου αφιερώσαμε λίγο περισσότερο χρόνο κατά την αξιολόγηση, οι περιοχές του στόχου 2 έχουν περιορισμένη κλίμακας ε, χρηματοδότηση, έχουν λιγότερο από 40 ευρώ κατά κεφαλή το χρόνο και εδώ βλέπουμε μεγάλη απόκληση και διαφορά σε σχέση με τα μεγάλης κλίμακας και χρονίζονται τα προβλήματα που έχουν ε, πολλές από αυτές τις περιοχές. Άρα θα πρέπει να δούμε πώς μπορούμε οι στατιστικές που έχουμε σε περιφερειακό επίπεδο να τις χρησιμοποιήσουμε για να, τις αξιο... για να αξιοποιηθούν σωστά. Βλέπουμε ταυτόχρονα όμως ότι ε, ότι έχουν ε, αυτές οι παρεμβάσεις καταλητικό ρόλο ως προς μια μακροχρόνια στρατηγική για την αναδιάρθρωση. Η αποτελεσματικότητα καταγράφεται στην ανάπτυξη Δηλαδή τα ποσοστά που επιτυγχάνονται τουλάχιστον δεν είναι χειρότερα από ό,τι σε περιφέρειες με λιγότερα προβλήματα. Όσον αφορά το μέλλον του στόχου 2. Πρώτη παρατήρηση, το όραμα και η δέσμευση των αρμόδιων για τη χάραξη της περιφερειακής πολιτικής είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ιδιαίτερα για, τους στόχους, για τις περιοχές του στόχου 2 και πολύ περισσότερο από το αρχικό, την αρχική δομή της εξειδίκευσης αυτής της περιοχής. Δηλαδή δεν έχει να κάνει μόνο με, την, ε, με τις επενδύσεις ή με την ιστορία της, ε, των ορχείων η ιστορία φερρυπίν ε, παραδοσιακά ναυπηγείων ή μικρών και μεσών επιχειρήσεων, μια περιφέρεια πέραν του ιστορικού της μπορεί να προχωρήσει, να ξεπεράσει, να κάνει την υπέρβαση αυτής της εξειδίκευσης και πάνω απ' όλα σημασία έχει το πόσο θα στρατευτούν σε αυτή την προσπάθεια αυτοί που είναι αρμόδια για τη χάραξη πολιτικής. Επίσης, Πολύ καλύτερα είναι τα αποτελέσματα όταν έχουμε συντονισμό του στόχου 2 και των περιφερειακών στρατηγικών. Αυτό προκύπτει ξεκάθαρα και από τις αξιολογήσεις και ορισμένες φορές οι ανταλλαγές εμπειριών ε, γίνονται μέσα από την ε, κοινοτική πρωτοβουλία Ιντερεκ. ενώ λησμονούμε μερικές φορές τη γνώση, την εμπειρία, την πείρα, τις ε, διδαχές που μπορούμε να αποκομίσουμε από τους στόχους 1 και 2. Χρειαζόμαστε περισσότερα στοιχεία σε σχέση με το στόχο 2, ιδιαίτερα ως προς τα μέτρα όχι στήριξη επιχειρήσεων τόσο όσο ε, επενδύσεων για την κοινωνική και την αδερφική συνοχή και αυτό διότι ήταν σαφές ότι στις ε, περιοχές Ανταγωνιστικότητα και απασχόληση. Υπάρχουν όντω περιφέρειες οι οποίε επιδιώκουν όχι μόνο την ανταγωνιστικότητα αλλά την εδαφική και κοινωνική συνοχή, δεδομένο το οποίο φαίνεται ότι δεν είχε καταγραφεί επαρκώ από του αρμόδιους για τη χαράξη πολιτική Και για να προχωρήσω στην τελευταία ή πρώτη τελευταία διαφάνεια, στα συστήματα διαχείριση και υλοποίηση που σα είχα παρουσιάσει και την προηγούμενη φορά, είναι όμω πολύ σημαντικά. να επισημάνω ότι οι χώρες, ε, η Ευρώπη των 10 ε, δεν είχαν επαρκή χρόνο βέβαια για την εφαρμογή προγραμμάτων, είχαν και περιορισμένη εμπειρία, αλλά τα αποτελέσματά του είναι πολύ καλύτερα από ό,τι αρχικά είχε προβλεφθεί, γιατί ήταν πολλέ πολλές που είχαν ακουστεί στο παρελθόν. Ε, δεν υλοποιήθηκαν φόβοι απορρόφησης, δυσκολιών απορρόφησης. Ε, υπάρχουν βέβαια κάποιες δυσκολίε που θα πρέπει να βελτιωθούν. και αυτό έχει να κάνει και με την Ευρώπη των 10 και με την Ευρώπη των 15, ότι στόχος είναι περισσότερο οι διαδικασίες και ο δημοσιονομικός έλεγχος, ε, έλεγχος που θα πρέπει να δώσουμε περισσότερη έμφαση και όχι αποτελέσματα των προγραμμάτων και αποτελεσματικότητας. Και επίσης δεν υπάρχει επαρκής αξιολόγηση ή υποστήριξη καλύτερα τη αξιολόγηση από του δείκτε. Ε, σε αυτά τα θέματα πρέπει να επανέλθουμε όταν έρθει η ώρα να διατυπώσουμε προτάσει για το μέλλον για να έχουμε πολιτική πιο εστιασμένη στα αποτελέσματα και λιγότερο στο πού πάνε τα χρήματα. Γιατί εμεί βεβαίω στην ομάδα πρέπει να σα πω ότι αισθανόμαστε μεγάλη δυσφορία όταν ε, κάποιοι έρχονται και μα λένε Α, τι καλά, καταφέραμε να δαπανίσουμε όλα τα λεφτά που έχουμε στη διάθεσή μα. Δεν είναι αυτό ο στόχο. Συνέπεια για μελλοντική πολιτική. Έχουμε πολλούς στόχους κοινωνικούς, περιβαλλοντικούς, οικονομικούς. Αυτό βλέπουμε ως ε, στοιχείο ισχύω της πολιτικής μας και όχι αδυναμίας. Πρέπει βεβαίω να το καταγράψουμε στο σχεδιασμό, την εφαρμογή και την αξιολόγηση. Δεν πρέπει να λησμονήσουμε τους περιβαλλοντικούς και κοινωνικούς στόχους να συζητούμε του οικονομικού στόχου. Και χρειαζόμαστε και προσδορισμό προτεραιοτήτων για τους διαφορούς στόχους σαφή προσδιορισμό προτεραιοτήτων, κατά το σχεδιασμό των προγραμμάτων και βέβαια χρειαζόμαστε και δείκτε. Επίση πιστεύουμε ότι χρειάζεται συγκέντρωση χρηματοδότηση στην κάθε περιφέρεια, χωρί αυτό να σημαίνει ότι θα πρέπει να υπάρξει ποικιλία στόχων, αλλά ταυτόχρονα πρέπει να υπάρχει συγκέντρωση της χρηματοδότησης με περιορισμένους ε, τομείς, ώστε να έχουμε την κρίσιμη μάζα και όχι μόνο βέβαια ένα στόχο. Τα μέτρα πολιτική δεν μπορούν να προσδοριστούν εκ των προτέρων. Πρέπει δηλαδή να ε, ευθυγραμμίζονται στις ανάγκες της περιφέρειας. Η αξιολόγηση μας λέει ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό οι ίδιες οι περιφέρειες να προσδιορίζουν ποιε είναι οι ανάγκες τους, ποιοι είναι οι στόχοι τους, που ε, θέλουν ε, να αναπτυχθούν τα μέσα πολιτικής, τα μέτρα πολιτικής, αλλά φέβαια θέλουμε να είμαστε και κάπως πιο για το μέλλον και έτσι ο καθένας θα πρέπει να γνωρίζει ποιοι είναι οι στόχοι για την πολιτική που θέλει και πώς θα αξιολογηθεί η επιτυχία του. Γιατί στο παρελθόν είχαμε μέτρο Πολιτική είχαμε χρηματοδότηση και μετά επαναρχόμασταν για να ρωτήσουμε τους ανθρώπους αν τα καταφέρανε, Του λέγαμε τα καταφέρατε, ήσασταν επιτυχεί και δεν είχαν απάντηση γιατί δεν ήξεραν καλά καλά τι θέλουν να αλλάξουν, τι θέλουν να μεταβάλουν και δεν υπήρχε συγκεκριμένο στόχος να επιτευχθεί. Πώς θα ξέρουμε λοιπόν αν είναι καλός ο στόχος και ανεξαρτήτως των επιλογών πρέπει αυτές να είναι δικαιολογημένες, αιτιολογημένες με βάση τις στρατηγικές Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Έτσι λοιπόν για να συνοψίσω, η αξιολόγηση αποδεικνύει συμβολή του Φεντέρος προς τη μείωση των αποκλήσεων. Η Ευρώπη των 25 στο σύνολό της κερδίζει χάρη στην πολιτική συνοχής Έχουμε περισσότερες γνώσει τώρα για το τι προσέφερε η πολιτική αυτή στους κύριου τομείς πολιτική μεταφορέ περιβάλλον και στήριξη επιχειρήσεων. Μπορούμε να αποδείξουμε ότι η πολιτική προσφέρει περισσότερο από απλή ανάπτυξη, καλύτερο περιβάλλον και κοινωνικά ωφέλη. Επίση, μπορούμε καλύτερα ακόμα να αξιολογήσουμε, αλλά τα ερωτήματα που καλούμε στα οποία καλούμε να δώσουμε απαντήσει είναι όλο και περισσότερα. Ξέρουμε περισσότερα, αλλά αυτό σημαίνει ότι γνωρίζουμε περισσότερο πόσα πράγματα δεν ξέρουμε. Ε, πολλά στοιχεία όμως ακόμα θα παρουσιαστούν σύντομα. Θα δημοσιεύσουμε τις ε, ε, αξιολογήσεις Urban και Interreg αυτό το μήνα. Για το ΙΣΠΑ θα έχουμε στα, τέλη του, στα μέσα του επόμενου χρόνου, ήδη όμως από φέτος θα έχουμε κάποια στοιχεία. Και επίσης σύντομα θα έχουμε ένα νέο δίκτυο εμπειρογνωμόνων που συνδυάζει τα στοιχεία για τις επιδόσεις 2007-2013, από τα προγράμματα δηλαδή αντίστοιχα για το κάθε κράτος μέλος και έτσι θα έχουμε πρώτα αποτελέσματα του 2011, στις αρχές του 2011, άρα βλέπουμε ότι έχουμε καλά αποτελέσματα, πιστεύω καλή αρχή έχουμε κάνει, χωρίς να επαρκούν αυτά που έχουμε δει μέχρι τώρα. Πάντως πρέπει να ενθαρρύνουμε τα κράτη-μέλη και κυρίως τις περιφέρειες να προβαίνουν σε προσθέσεις αξιολογήσεις έτσι ώστε να αναπτυχθεί αυτό το κόρπους των στοιχείων, γιατί δεν υπάρχει επαρκής αξιολόγηση ε, δεν υπάρχει αξιολόγηση η οποία να δίνει απαντήσει σε κάθε ερωτηματικό. Εάν όμως έχουμε αρκετό αριθμό αξιολογήσεων, σε τακτικούς ρυθμούς, με, με καλά στοιχεία, τότε αυτά τα αποτελέσματα μπορούμε να τα αξιοποιήσουμε για να ε, κάνουμε επιλογές για νέες πολιτικές εφόσον κρυθεί αυτό απαραίτητο. Ε, I think I can say on Νομίζω ότι μπορώ να πω εκ μέρους των συναδέλφων. Ήταν πάρα πολύ χρήσιμη αυτή η παρουσίαση. Ε, και πολύ χρήσιμη για την συζήτηση που θα ακολουθήσει τώρα. Ο πρώτος είναι ο κύριος Πίπερ που έχει γραφεί στο κατάλογο των αγορητών. Μάρκος, έχεις το λόγο. Σας ευχαριστώ. Ο κύριος Άνερ και η κυρία Γκαφέ μας έκαναν πολύ διεξοδικές και ακριβείς αναλύσεις. Έχω κάποιες ερωτήσεις που σχετίζονται και με την επόμενη περίοδο. Ποια ήταν η εμπειρία σας σε ό,τι αφορά την χρησιμοποίηση του Ταμείου Συνοχής και του Περιφερειακού Ταμείου. Υπάρχει υπερβολικά γραφειοκρατική συνύπαρξη μεταξύ των δύο ταμείων. Μιλήσατε για μια συνοπτική εργασία που έγινε, αλλά μήπως είναι περίπλοκα τα πράγματα. Μήπως το Ταμείο συνοχή και το Περιφερειακό Ταμείο θα πρέπει να συγχωνευτούν τελικά, μήπως αυτό είναι το καλύτερο συμπέρασμα και για λόγους αποτελεσματικότητας, ενίσχυσης της αποδοτικότητάς τους. Αυτή την απόρρεια έχω. Και θα ήθελα κύριε Άνερ να μου απαντήσετε. Έστω και γενικά. Μία χώρα σαν την Ελλάδα μεταξύ του 2000 και του 2006 ήταν μια χώρα που παραβίασε το Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης. Και εκεί, αντί να μειωθούν οι ανισότητες, ενισχύθηκαν. Μου είπατε ως δικαιολόγηση την ε, ανάπτυξη της Αθήνας. Αλλά αυτή η χώρα επανειλημμένως παραβίασε τα, στοιχεία, τα κριτήρια της σταθερότητας. Μπορούμε λοιπόν να είμαστε βέβαιοι ότι τα κονδύλια που δίνονται στις χώρες αυτές αξιοποιούνται δεόντως. Υπάρχουν κατάλληλοι μηχανισμοί ελέγχου, για τη χρησιμοποίηση αυτών των κονδυλίων. Και είναι και πολύ επίκαιρο αυτό το θέμα. Γιατί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν χρησιμοποίησε το κατάλληλο άρθρο του Ταμείου Συνοχής. που προβλέπει ότι όταν μια χώρα παραβιάζει τις διατάξεις αποκλείεται από την παροχή των κονδυλίων της συνοχής. Γιατί δεν συνέβη κάτι τέτοιο, γιατί δεν ε, εφάρμοσε η Επιτροπή το σχετικό άρθρο. Είναι πολύ συγκεκριμένη η ερώτηση. Έχω και μια άλλη ερώτηση για το μέλλον της πολιτικής συνοχής. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα χρησιμοποιήσει έναν αυτοματισμό σε ό,τι αφορά τα, τις χώρες που συστηματικά παραβιάζουν τα κριτήρια της σταθερότητας. Και για τις χώρες που δημιουργούν μεγάλα προβλήματα υπάρχει δυνατότητα αυτόματης εφαρμογής κυρώσεων σε περίπτωση που παραβιάζονται τα διαρθρωτικά ταμεία. Επίσης, στην Ένωση των 15 μπορούμε να έχει νόημα να, χρησιμο, να χρηματοδοτούμε την α, ε, κατασκευή αυτοκινητοδρόμων. Και αν αυτό αναπτύσσει την αγορά των ανατολικών χωρών, ίσως θα μπορούσαν να χρηματοδοτηθούν οι διασυνδέσεις με τις δυτικές χώρες. Κάτι τέτοιο θα ωφελήσει και τις χώρες Ανατολικής Ευρώπης. Εγώ πιστεύω ότι θα πρέπει να εξακολουθούμε να χρηματοδοτούμε κατασκευή αυτοκινητοδρόμων, γιατί κάτι τέτοιο ευνοεί την ανάπτυξη των διαφόρων περιοχών. Κυρία Ουκασεύσκα. Κυρία Πρόεδρε, εγώ δεν έχω καμία αμφιβολία ότι το Ταμείο Συνοχή ήταν πολύ επιτυχημένο. Μπορεί να μην ήταν τόσο επιτυχημένο όσο φιλοδοξούσαμε και περιμέναμε, πάντω σίγουρα η επιρροή του στην υλοποίηση των συγκεκριμένων στόχων ήταν πολύ σημαντική. Έχω μία ερώτηση. Αν είναι δυνατόν να γίνει η αξιολόγηση και η απομονωμένη επιρροή της, ε, του Ταμείου Συνοχής στην ανάπτυξη των περιοχών, ανεξάρτητα δηλαδή από την επιρροή άλλων ε, ταμείων και πολιτικών. Επίσης, ε, πιστεύετε ότι μπορούν να χρησιμοποιηθούν οι μέθοδοι του μάρκετινγκ για να προωθηθούν τα προγράμματα της πολιτικής συνοχής και να βελτιωθεί επικοινωνιακά το η εικόνα της, ε, της περιφερειακής πολιτικής, γιατί γίνονται τεράστιες προσπάθειες, αλλά δεν ξέρει ο κόσμος ότι πολλές τέτοιες προσπάθειες χρηματοδοτούνται από κοινοτικά κονδύλια. Ίσως εκεί θα πρέπει να καταβάλουμε μια επικοινωνιακή προσπάθεια, χρησιμοποιώντας ακόμη και μεθόδους marketing για την προβολή αυτής της πολιτικής. Θα ήθελα επίσης να ρωτήσω αν εξετάσατε την ε, πρόσβαση στα κοινοτικά κονδύλια συγκεκριμένων χωρών, μεμονωμένων χωρών. Γιατί ο κύριος Πιπέρα αναφέρθηκε στην υπερβολική γραφειοκρατία. Η Ευρωπαϊκή Ένωση όμως είναι μία και μόνη, οπότε η πρόσβαση θα πρέπει να είναι αντίστοιχη σε όλες τις ε, χώρες μέλη. Έχω την αίσθηση όμως ότι η πρόσβαση αυτή στα κοινοτικά κονδύλια σε ορισμένες χώρες είναι πολύ εύκολη, ενώ σε άλλες είναι ολόκληρος γολγοθάς για να φτάσουν στα κοινοτικά κονδύλια. Υπάρχουν πολλοί γραφειοκρατικές διαδικασίες, μία σωρία που θα πρέπει να ε, πραγματοποιούν οι ενδιαφερόμενοι προκειμένου να φτάσουν στα κοινοτικά κονδύλια και ούτω καθεξής. ευχαριστώ πολύ και μου επιτρέπετε πρώτα να δώσω απαντήσει στον κύριο Πίπερ εμπειρία από το Ταμείο Συνοχής και το Περιφερειακό Ταμείο. Ναι, το όντι ήταν περίπλοκη κατάσταση στο παρελθόν, διότι το Περιφερειακό Ταμείο είχε μια διαδικασία προγραμματικού σχεδιασμού, ενώ το Ταμείο Συνοχής δούλευε με συγκεκριμένα σχέδια, project. Για την περίοδο 2007-2013 όμως, το Ταμείο Συνοχής με τα σχέδιά του, τα, τα σχέδια μάλλον ενσωματώθηκαν στα περιφερειακά προγράμματα των κρατών και έτσι προχωρήσαμε πιστεύω, ε, πραγματοποιήσαμε ένα βήμα πρόοδου. Πλην όμως παραμένει ακόμη ε, αρκετή, αρκετός βαθμός επικάλυψης, για να μην πω και αντιφάσεων μεταξύ των δύο αυτών παρεμβάσεων, αυτών παρέμβασης. Φερρυπίν, ένα μεγάλο σχέδιο από το Ταμείο Συνοχής μπορεί να, προσδιορίζεται διαφορετικά ε, στο Ταμείο το περιφερειακό, δηλαδή το μεγάλο σχέδιο να μην έχει τον ίδιο ορισμό στο περιφερειακό ταμείο. Και νομίζω ότι βρισκόμαστε σε ένα στάδιο τώρα που και τα δύο ταμεία θα πρέπει να έχουν τους ίδιους κανόνες, θα πρέπει να ισχύουν οι ίδιοι κανόνες για τα δύο ταμεία. Τώρα, εάν πρέπει να προχωρήσουμε και περαιτέρω, αυτό είναι πολιτικό όμως ερώτημα, εάν πρέπει να προχωρήσουμε περαιτέρω για να πούμε καταργούμε το Ταμείο Συνοχής και το συγχωνεύουμε μέσα σε μια μεγάλη περιφερειακή πολιτική που καλύπτει και τη συνοχή και τις περιφέρειες είναι ένα δύσκολο ερώτημα. Εάν όμως στο προσεχές βήμα τώρα πούμε τουλάχιστον ότι για την εφαρμογή των δύο ταμείων ισχύουν για το ίδιο πρόγραμμα ακριβώς οι ίδιοι κανόνες ή μη τι άλλο έχει πραγματοποιηθεί σημαντικό βήμα προόδου και βέβαια από εκεί και πέρα λαμβάνεται η πολιτική απόφαση ε, εάν θέλει κανείς να πει ότι χρειάζονται για να χορηγηθούν τα υποστώσεις δύο διαφορετικά ταμεία ή αν μπορούμε να μιλήσουμε για ένα ταμείο. Τώρα, για την Ελλάδα και το Ταμείο Συνοχής. Το όντι οι περιφερειακές αποκλίσεις, διαφορές μέσα στην Ελλάδα όντως έχουν ενισχυθεί. Πράγμα το οποίο νομίζω μπορεί να εξηγηθεί από την ραγδαία ανάπτυξη ιδιαίτερα της Αθήνας στην τελευταία περίοδο. Αυτό με απασχόλησε βέβαια και σε σχέση με τα μακροοικονομικά προβλήματα της Ελλάδας μας απασχόλησε το πώς στο μέλλον τέτοιου είδου ζητήματα στον τομέα της πολιτικής συνοχής μπορούν να βρούνε κάποια ανταπόκριση. Πώς θα αντιδρούμε. Στο πρώτο σημείο που θα θέλω να, το οποίο θέλω να καταστήσω σαφές είναι ότι δεν μπορούμε να έχουμε ανάπτυξη βιώσιμη αν δεν υπάρχουν δεδομένα, αν δεν υπάρχει πλαίσιο σταθερό, μακροοικονομικό. Δηλαδή και τα δύο πρέπει να είναι αλληλένδετα δεν μπορούμε να τα ξεχωρίσουμε το ένα από το άλλο. Στη δε περίπτωση της Ελλάδας ε, μας απασχόλησε το κατά πόσον για τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο το Ταμείο συνοχή θα μπορούσε να αξιοποιηθεί για να γίνει πρόταση προς, τους, ε, προς το Συμβούλιο των Υπουργών να αξιοποιηθεί το Ταμείο Συνοχής υπέρ της Ελλάδας. Καταλήξαμε όμως το συμπέρασμα ότι για την Ελλάδα το μόνο το οποίο σήμερα θα μπορούσε ως στήριξη να βοηθήσει για την επανεκκίνηση της οικονομικής ανάπτυξης θα ήταν τα κονδύλια του Ταμείου Συνοχής. Του Διαρθρωτικού Συνόμου Ταμείου. Και αυτό ήταν ακριβώς το ζήτημα το οποίο μας απασχόλησε περισσότερο. Και δεν θα σας κρύψω βεβαίως, σε σχέση με το μέλλον μας απασχόλησε ήταν το θέμα αυτό, μαζί με τους συναδέλφους Γενικής Διεύθυνσης που ασχολούνται με τα θέματα τα οικονομικά και τα νομισματικά. Μας απασχόλησε λοιπόν το πώς θα μπορούσαμε ενδεχομένω να έχουμε μια πιο συστηματική, ένα πιο συστηματικό προσδιορισμό όρων για την διάθεση των κονδυλίων των, του Διευθυντικού Ταμείου και των όρων ε, της ε, μακροοικονομικής σταθερότητας. Για μας αυτοί οι όροι, οι προϋποθέσεις θα μπορούσαν να προσδιοριστούν σε τρία διαφορετικά επίπεδα. Το πρώτο, όπως είπα, μακροοικονομική σταθερότητα, με κύριο ερώτημα, εάν θέλουμε τα πράγματα να τα αφήσουμε όπως έχουν τώρα, δηλαδή Ταμείο Συνοχής και δυνατότητα με πρόταση της Επιτροπής Ταμείου Συνοχής και με απόφαση βέβαια του Συμβουλίου να τεθεί σε λειτουργία, να ενεργοποιηθεί. Εάν θα πρέπει αυτή η δυνατότητα που έχουμε για το Ταμείο Συνοχή να επεκταθεί σε, όλο, σε όλα τα διευθυντικά ταμεία και αν πρέπει αυτή την απόφαση να την ε, συνδυάσουμε με μια αυτόματη θέση σε λειτουργία Τη στιγμή δηλαδή όπου έχει φτάσει ένα σημείο συγκεκριμένο διαδικασία της ε, σταθεροποίησης, να λέμε stop, εδώ έρχεται μέχρι ότου να υπάρχει, εδώ σταματάνε τα πάντα μέχρι ότου έρχεται μια αξιόπιστη πρόταση, ένα σχέδιο αξιόπιστο. Όλα αυτά τα έχουμε ε, συζητήσει, δεν έχουμε καταλήξει όμως παρά μόνο στο να πούμε ότι δυνητικά θα υπήρχε αυτή η δυνατότητα στο μέλλον. Πάντως σίγουρα ένα σημείο το οποίο μας απασχολεί. Ένα άλλο σημείο το οποίο μας απασχολεί, οι ε, προϋποθέσεις, είναι το πώς θα συνδυάσουμε καλύτερα στο μέλλον ή θα συσχετίσουμε καλύτερα αφενός με τα εθνικά προγράμματα μεταρρύθμισης που αναπτύσσονται και στο πλαίσιο του Ευρώπη 2020 πρέπει να αναπτυχθούν καλύτερα και αφετέρου το διαρθρωτικό τα διαρθρωτικά ταμεία. Δηλαδή, για να το πω καλύτερα, Πώς θα βεβαιούμαστε ότι τα διαρθρωτικά ταμεία αξιοποιούνται για τα μεταλαφμιστικά αυτά προγράμματα, για την απασχόληση κτλ. κατά τρόπο αποτελεσματικό. Αγορά εργασίας και νομίζω υπάρχει και μια πρόταση, δεν ξέρω αν την έχετε δει κι εσείς, μια πρόταση του καθηγητή κ. Μόντι, κατά την υλοποίηση της εσωτερικής αγοράς να υπάρχει ένα είδος αποθεματικού στο οποίο θα λέμε ότι ένα μικρό ποσοστό των πιστώσεων των αθλητικών ταμείων δεσμεύονται εκεί και αποδεσμεύονται μόνο όταν ένα κράτος έχει φτάσει να εκπληρώσει τις συγκεκριμένες προϋποθέσεις ε, ολοκλήρωσης της εσωτερικής αγοράς. Πολλέ ιδέες έχουν εκφραστεί στην υπόθεση αυτή, ε, ιδέες οι οποίες πρέπει να συζητηθούν με προσοχή, να εξεταστούν με προσοχή, ιδέες οι οποίες εν τέλει μπορεί να οδηγήσουν σε πολύ σημαντικές πολιτικές αποφάσεις. Και σας διαβεβαιώ δεν είναι ζήτημα καθόλου τεχνοκρατικό αυτό. Είναι ζήτημα πολιτικών επιλογών. Απλώς πρέπει να ξέρετε κι εσείς ότι και από την πλευρά μας τα μελετούμε όλα αυτά τα πράγματα και εξετάζουμε το πώς στην πράξη θα μπορούσαν ενδεχομένως αν ληφθεί η απόφαση να ε, ε, εφαρμοστούν όλα αυτά. Για δε την παρατήρηση, α ναι, αν μου επιτρέπετε λοιπόν τώρα για το τελευταίο επίπεδο, το τελευταίο, το τρίτο επίπεδο, το οποίο μας ενδιαφέρει ιδιαίτερο σε εμά στον τομέα της ε, διαφορετικής πολιτικής, είναι το πώς στο μέλλον θα εξασφαλίσουμε ε, μια σαφέστερη συμμετοχή μας ε, ή σε αυτή τη δουλειά αν θέλετε της ε, εποπτείας, της επιτήρησης που κάνουμε με περισσότερη αξιοπιστία, πιο καλή αποδοτικότητα της δουλειάς που γίνεται επί τόπου. Έτσι ώστε να μην υπάρχει τόσο, να μην δίνεται μεγάλο βάρος στους λεπτομερείς μηχανισμούς, γραφειοκρατικούς μηχανισμούς, μηχανισμούς μετρήσεων ε, πώς μπορούμε δηλαδή πιο καλά να κάνουμε τις μετρήσεις εν ολίγης. Τα τρία επίπεδα όπως είπα, μακροοικονομική σταθερότητα, συσχετισμός με τα μεταρρυθμιστικά προγράμματα και βάση της δουλειάς για μας πώς θα έχουμε τη βεβαιότητα ότι σε μια περίοδο μάλιστα που είναι όλο και λιγότερα τα διαθέσιμα κονδύλια, αυτά τα οποία διαθέτει η διαρθρωτική πολιτική πηγαίνουν στις πραγματικά απαραίτητες και χρήσιμες επενδύσεις και τα αντίστοιχα σχέδια. Επόμενη ερώτηση. Ο αντίκτυπος της πολιτικής συνοχής μπορεί να απομονωθεί μέσα σε μια ε, σχέση αιτιότητας η απάντηση είναι όχι, τουλάχιστον με την απλή παρατήρηση στατιστικών δεδομένων, δηλαδή θα πρέπει να προχωρήσουμε σε μια πολύ πιο περίπλοκη ανάλυση μοντέλου και κάθε φορά αυτό σημαίνει επιπλέον προβλήματα πρέπει να σας πω, η κάθε ανάλυση, το κάθε μοντέλο έχει δικά του ε, προβλήματα και ελλείψεις Ταυτόχρονα δηλαδή χρησιμοποιούν δεδομένα διαφορετικών προελεύσεων τα μοντέλα αυτά και εμεί προσπαθούμε βλέποντα διαφορετικά μοντέλα με τα διαφορετικά στοιχεία που χρησιμοποιούν αυτά να καταλήξουμε σε μια διαπίστωση. Εάν δούμε δηλαδή ότι πολλά μοντέλα μα δίνουν το ίδιο, το ίδιο αποτελέσματα κάθε φορά, τότε ναι μπορούμε να τα θεωρήσουμε αξιόπιστα και τα αποτελέσματά του αυτά φυσικά. Και επίση θα ήθελα να σα πω ότι, εκτό γνωρίζω εγώ, αλλά η Βερόνικα θα μα δώσει περισσότερε πληροφορίε, ότι Λιγότερε είναι οι πληροφορίε που έχουμε στη θέση μα, οι συγκρίσιμε πληροφορίε που έχουμε στη θέση μα, που μα επιτρέπουν να φτάσουμε σε ανάλυση τη λεπτομέρεια για την πρόσβαση στα επιμέρου κονδύλια στο κάθε κράτο, αλλά η εμπειρία που έχουμε συλλέξει, έστω και αν δεν υπάρχει συστημική ανάλυση πίσω από αυτήν, η εμπειρία που έχουμε συλλέξει μα δίνει όντω μια ορθή εικόνα ω προ τον τρόπο με τον οποίο διαφορετικά κράτη ε, ε, έχουν αναπτύξει σε μεγαλύτερο ή μικρότερο βαθμό δυσκολίες ή γραφειοκρατικά προσκόμματα ως προς την πρόσβαση σε αυτά τα κονδύλια. Ή μερικές φορές βλέπουμε ότι είναι πιο δυσκίνητη η εθνική νομοθεσία για την πρόσβαση από ό,τι θα χρειαζόταν. Όπου έχουμε δει τέτοιου είδου περιπτώσει λοιπόν, σε συνεργασία με τι περιφέρειες και τα κράτη-μέλη, προσπαθούμε να του πείσουμε να απλουστεύσουν, να αλλάξουν την εθνική του νομοθεσία, τι διατάξει του. Και το πρόβλημα το οποίο διαπιστώνουμε πάντοτε είναι αυτό τη μέρημνα για το δημοσιονομικό έλεγχο τη Ευρωπαϊκή Ένωση, ότι δηλαδή όταν προσδιορίζεται ένας κανόνας, το επίπεδο στο οποίο στη συνέχεια αναπτύσσεται η δραστηριότητα, δηλαδή το περιφερειακό ή και το τοπικό ακόμη επίπεδο, θα πρέπει να έχει και τους αντίστοιχους κανόνες και πολλές φορές βλέπουμε ότι οι κανόνες αυτοί για την εφαρμογή είναι ακόμη πιο περίπλοκοι, διότι υπάρχει πάντα η ανησυχία μην έρθει ο έλεγχος από την Ευρωπαϊκή Ένωση και δεν είναι ικανοποιητικός. Δηλαδή μπορεί να έχουμε κάπου αντί για 100% τήρηση ή, ή διατάξεις περιτήρησης στις περιφέρειες ή το τοπικό ακόμα επίπεδο να έχουν φτάσει στο 140%. Χωρίς αυτό να σημαίνει πάντοτε ότι υπάρχει καλύτερη αποτελεσματικότητα. Ευχαριστώ πολύ. Αγαπητοί συνάδελφοι, έχουμε 11 γραμμένο στον κατάλογο. Παρακαλώ να είστε πιο σύντομοι. Η το Ευχαριστώ καταρχά. Και συγχαρητήρια. Πολύ καλή έκθεση. Στην αρχή όταν ε, το είδα στο πρόγραμμα είπα «Ε, καλά εντάξει. Έκθεση εκ των υστέρων, αξιολόγηση, ποτέ δεν είναι συναρπαστικά αυτά τα πράγματα κυρίω μα ενδιαφέρει τι πρόκειται να γίνει, αυτό τι έχει γίνει, αλλά η ανάλυση την οποία προέβηται, μπράβο, συγχαρητήρια, ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρουσα και συνερπαστική. Και πάνω απ' όλα μα δείχνει τι μπορούμε να διδαχθούμε από το παρελθόν, από την εφαρμογή μέχρι τώρα των προγραμμάτων. Θα ήθελα εκεί που λέτε ότι ενδεχομένως να μην υπάρχουν μετρήσιμα στοιχεία, να επισημάνω ότι χρειάζεται περισσότερη προσοχή και βεβαίως πάνω απ' όλα στη δημιουργία θέσεων εργασία, ε, πιο δύσκολο να προσμετρήσουμε τι θέσει εργασία που δημιουργούνται στι δημόσιε μεταφορέ σε σχέση με την κατασκευή νέων οδικών αρτηριών ή τι μπορεί να προσφέρει μια ε, πιο περιβαλλοντική πολιτική, στη, πολιτική στις περιφέρειες ως προς τις δημιουργία θέσεων εργασίας. Πρέπει όμως να επισημάνω ότι υπάρχει και έκθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου από την Επιτροπή Απασχόλησης ως αρμόδια κατουσίαν Επιτροπή με πολύ καλή συνεργασία και της Περιφερειακής Επιτροπής με την κυρία Βέστφαλ και νομίζω ότι στην Επιτροπή μας μπορούμε να έχουμε πολύ καλές ιδέες για το πόσες θέσεις εργασίας μπορούν να προκύψουν από την χρηματοδότηση αυτή. Γιατί τα βλέπουμε όχι μόνο από την οπτική γωνία της Επιτροπής, αλλά και από την εμπειρία που έχουμε από τα κράτη-μέλη μας όλα αυτά. Νομίζω μπορείτε να αξιοποιήσετε και αυτή την εμπειρία. Ε, δεύτερη ερώτηση, η παρατήρηση, γραφειοκρατία και έλεγχος, αυτό που μόλις είπε και ο κύριος Άνερ τώρα. Δηλαδή, ο φόβος να ενισχύεται διαρκώς η γραφειοκρατία, μετά να επιρρύπτονται οι ευθύνε για την ενισχυμένη γραφειοκρατία στην Ευρωπαϊκή Ένωση, έστω και αν δεν είναι αυτή η υπεύθυνη. Υπάρχει ένα σφάλμα όμω και βλέπω ότι ναι, μεν δεν εμφανίζεται στην έκθεσή σα τώρα, αλλά εν γέννη στην προηγούμενη έκθεση του 2007, 2007-2013, ίσω να έχει κάποια σημασία να το δούμε αυτό ότι δηλαδή ή επιτόπου έλογοι και ξέρουμε για ποιους λόγους, που διεξάγετε εσείς στις διάφορες περιφέρειες, στα κράτη-μέλη, έχουν μειωθεί. Γιατί λοιπόν να, να μειώνουμε τους ελέγχους και με ποια κριτήρια προσδιορίζονται ε, οι έλεγχοι, ε, ποιος μάλλον ορίζει τα κριτήρια με βάση του οποίους γίνονται οι έλεγχοι, πώς γίνεται αυτό και γιατί γίνεται αυτό, έχουν καταργηθεί σε θέσεις εργασία. έχουν οι περιοφέρειες αυτές αναπτυχθεί, ποιο θα το κρίνει αυτό και γι' αυτό νομίζω ότι θα ήταν καλό να υπάρχουν περισσότεροι επιτόπιοι έλεγχοι. Να μην λέμε δηλαδή ε, ότι αυτοί οι έλεγχοι επιτόπου είναι όπως ε, στο θεατρικό έργο του Γκογκόλ ο επιθεωρητής επιστρέφει, ε, ε, έρχεται, αλλά να μπορεί η Επιτροπή με τις επισκέψεις αυτές να διαπιστώνει που έχουν γίνει σφάλματα, τι μπορεί να διορθώσει ενδεχομένω με νέες διατάξεις, με την τροποποίηση των κανονισμών, που μπορεί να βοηθήσει μια περιφέρεια ή που, εν πάση περιπτώσει, έγκυται το πρόβλημα. Όταν λοιπόν έχετε χρησιμότητα ο επιτόπιος έλεγχος, το να μειώνονται οι επιτόπιοι έλεγχοι, ασφαλώς δεν μπορεί να είναι καλή επιλογή. Θέλουμε μεγαλύτερη συχνότητα. Και εμεί εδώ στην Επιτροπή μα οπωσδήποτε βλέπουμε ότι χωρί να ενισχύεται η γραφειοκρατία έχουμε καλύτερα αποτελέσματα. Γιατί πολλά πράγματα με την απευθεία επικοινωνία ρυθμίζονται. Αντί να έχει κανεί άγχο και φόβο για τον έλεγχο, βλέπει τον ε, συνομιλητή του και συζητά μαζί του. Ίσως δε μαζί με, το ταμείο, μαζί με το συνέδριο να συζητηθεί και να λέμε ας πάμε να κάνουμε μαζί την προληπτική αυτή ε, επίσκεψη Αντί να περιμένουμε να κλείσει ο προπολογισμό και η εκτέλεσή του και να έρχεται εκ των υστέρων το ελεκτικό συνέδριο για να επιστώσει που έχουν γίνει τα σφάλματα, α θέλει μαζί έναν εκπρόσωπο κατά τη διάρκεια τη εκτέλεση για να βεβαιούνται ότι πάνε καλά όλα. Εν πάση περιπτώσει, δοκιμαστικά, πειραματικά θα μπορούσαμε να το, να το δοκιμάσουμε αυτό. Και θα μπορούσατε να το συστήσετε με τα κρατημέλη και να πείτε ότι να, μαζί με το ελεκτικό συνέδριο θα ερχόμαστε για να βλέπουμε πώς προχωρεί η εκτέλεση των κονδυλιών αυτών και βέβαια έτσι ασφαλώς περιορίζουμε την γραφειοκρατία. Και τελευταία παρατήρηση. Είπατε ότι θέλετε να έχετε απευθείας ε, εξέταση των εθνικών μεταρρυθμιστικών προγραμμάτων. Ναι, αλλά μήπω εδώ λησμονείται η σημασία των περιφερειών, γιατί εδώ αυτό μα ενδιαφέρει εμά. Τα εθνικά προγράμματα μεταρρύθμιση δεν στρέφονται παρετά προ την υποστήριξη των ε, περιφερειών. Και εάν τα κοιτάζετε αυτά, τελικά θα κοιτάτε μόνο τι έχει αποφασίσει το το επίπεδο, το κεντρικό επίπεδο. Η έκθεση Πάκα είχε πει ότι η αποτελεσματικότητα σημαίνει να βοηθούμε στην ανάπτυξη των περιφερειών, όχι μόνο του κεντρικού επίπεδου, του εθνικού επίπεδου. Και επιπλέον η συνοχή προς αυτό το στόχο πρέπει να, να πηγαίνει. Ευχαριστώ κύριε Σωρό. Ε, Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Μια απλή ερώτηση. Στην κυρία Διευθύντρια της Μονάδας Αξιολόγησης. η αξιολόγηση που κάνατε αφορά επίσης τα κονδύλια που δίνονται στις ε, ε, περιφέρειες που βρίσκονται στην εξωτερική περιφέρεια της Ένωσης και στην περίπτωση αυτή είναι δυνατό να αφαιρέσετε από την συνολική αξιολόγηση τα κονδύλια και τις μελέτες που αφορούν αυτές τις ε, ε υπερπεριφερειακές περιοχές. Επόμενος μιλητής, Ο κύριος Κύριλοφ. Ευχαριστώ. Καταρχήν σας συγχαίρω κύριε Άνερ και κυρία Γκάφε για την υψηλό επίπεδο παρουσίαση που μας κάνατε. Θα μπορούσα να φέρω κάτι που είπε ε, ένας διάσημος καλλιτέχνης είπε μην φοβάτε την τελειότητα, ποτέ δεν μπορείτε, θα μπορέσετε να την πετύχετε. Σχεδόν αυτό πετύχατε όμως. Δηλαδή, μας δώσατε πολλά στοιχεία γνώσεων και πληροφόρησης αρκετά πολεμοφόδια αυτή τη στιγμή να υποστηρίξουμε τον κεντρικό άξονα της πολιτικής συνοχής. Αυτό είναι σημαντικό και για όλη την Ένωση. Όλα τα στοιχεία υποστηρίζουν την κατεύθυνση αυτή. Στην κρίσιμη περίοδο που ζούμε όσον αφορά την οικονομία και τα χρηματοπιστωτικά, γιατί όλοι το νιώθουμε αυτό στις χώρες μας, και αυτό που θέλω να πω είναι θα έπρεπε ενδεχομένως να δούμε το, τι συμβαίνει σήμερα, πόσο γρήγορα μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε αυτά τα κονδύλια η απλούστευση πρέπει να αρχίσει γρήγορα. Μερικές χώρες χρειάζονται βοήθεια. Από ό,τι φαίνεται περιμένετε χειρότερα πράγματα από τις ε, νέες χώρες όσον αφορά την απορροφητικότητα. Ωστόσο, έχουμε ακόμα δυσκολίες. Στη χώρα μου, πρόσφατα, μια επιστολή του Γενικού Διευθυντή δημοσιεύτηκε ζητούσε από τις αρχές να επιταχύνουν τις προσπάθειές τους και σας συγχαίρω γι' αυτό. Θα ήθελα κύριε Άνερ να μας πείτε, όχι συγκεκριμένες χώρες, αλλά μας πείτε πόσες χώρες χρειάζονται τέτοιου είδους πίεση αυτή τη στιγμή, γιατί βρισκόμαστε σε κρίσιμη φάση. Υπάρχει ακόμα χρόνος να έχουμε καλή χρήση των κονδυλίων που υπάρχουν. και να συνεργαστούμε και με τους συναδέλφους στα εθνικά κοινοβούλια. Γιατί το να τις χώρες για πιο αποδοτική χρήση των κονδυλίων να τα προγράμματά τους γκέρους, όλα αυτά είναι χρήσιμα. Αναφερθήκατε σε, στα ελληνικά προγράμματα για τις μεταφορές που είναι σημαντικές όχι μόνο για μία χώρα αλλά και για την διασυνοριακή συνεργασία περισσότερων χωρών γενικότερα. Τι θέλω να πω. Σας συγχαίρω επιδοκιμάζω αυτά που είπατε. Τέτοιου είδου μελέτες και αναφορές μας βοηθάνε να μειώσουμε στο μέλλον πειρασμούς γραφειοκρατικής φύσης. Γιατί ξέρουμε προς τα που πάμε και ξέρουμε να αποφύγουμε περιττή γραφειοκρατία. Ο συνάδελφος Λάμπερ Φανίνης δρόμο. Ευχαριστώ πολύ. Και εγώ σας συγχαίρω για την πάρα πολύ ενδιαφέρουσα αυτή μελέτη. Ωστόσο, έχω κάπως την εντύπωση ότι είναι ωραία αυτά τα αποτελέσματα. Και ένα ευρώ που το έχουμε στη τσέπη μπορούμε να το δαπανίσουμε μία φορά. Έχουμε αυτό το μοντέλο που φαίνεται ότι λειτουργεί καλά. Αύξησε το ΑΕΠ κατά 2% από το 2000 μέχρι το 2006. Χθε ήμουν στην Επιτροπή Ήτρα και ήρθε η Επίτροπος Κρούς και μας παρουσίασε την πολιτική της για τα επόμενα χρόνια. Μας παρουσίασε ε, μια πλαστική κάρτα, είπε αυτή θα την έχουν όλοι. Ωραία, αλλά πώς θα το πετύχει αυτό δεν ξέρω. Εμείς εδώ Έχουμε νούμερα και γεγονότα, αλλά δεν συμφωνούμε για το μοντέλο ακόμα. Δεν έχουμε συμφωνήσει. Και είναι επικίνδυνο αυτό. Έρχεται η κυρία Κρούς και λέει όλοι να έχουμε ένα είδος πλαστική κάρτα σαν την πιστοτική κάρτα ας πούμε όλοι. Αν επενδύουμε ένα ευρώ στις περιοχές στόχου 2 εγώ λέω πρέπει να υπάρχει, ότι πρέπει να υπάρχει ένα συγκεκριμένο μοντέλο. Αν ο νέος δημοσιονομικός κανονισμός με την αναθεώρησή του θα απαιτεί περισσότερους ελέγχους ή θα απαιτεί περισσότερη ελευθερία και εμπιστοσύνη. Αν τα κράτη-μέλη των συγκεκριμένων στόχων αναλαμβάνουν την οικονομική ευθύνη για να το κάνουν, καλό. Αν όχι όμως, Αν όχι όμως, τι θα κάνουμε. θα ζούμε στον 20ο αιώνα, θα στηριζόμαστε μόνο στους ελέγχους, αν έχουμε στόχους, αν έχουμε τη στρατηγική Ευρώπη 2020 για μια πιο βιώσιμη και πράσινη Ευρώπη. Ας δούμε ότι ναι μεν χρειάζεται η ευρωπαϊκή χρηματοδότηση, χρειάζεται όμως και συνευθύνη και συγχρηματοδότηση από τα κράτη-μέλη αν δαπανάμε μόνο κοινοτικά κονδύλια, ευρωπαϊκά κονδύλια και μετά συζητάμε τα διάφορα μοντέλα και διάφορες μελέτες, στο σύστημα αυτό που λειτουργεί με 17 χώρες θα κινείται όλο και με μεγαλύτερη βραδύτητα. Έχουμε δηλαδή ένα σύστημα που δεν μας επιτρέπει να ελέγχουμε τα πάντα και δεν είναι μια πάρα πάρα πολύ θετική εικόνα. Και νομίζω ότι ο κύριος Φίπερ έχει δίκιο όταν λέει ότι είναι υποχρέωση των κρατών μελών και μετά πλέον έχουμε τις παρεμβάσεις των διαφορών ταμείων μετά. Εσείς μελετήσατε την περίοδο 2000-2006. Πάει πέρασε αυτό. Θα μπορούσατε να μας δώσετε και πιο συγκεκριμένα νούμερα και δεδομένα. Γιατί όταν πάμε να ορίσουμε προτεραιότητες και πού θα επενδύσουμε και πώς σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, χρησιμοποιούμε κονδύλια για ανάκαμψη της οικονομίας εμείς στο ΕΛΚ κάναμε μία ακρόαση για τους νέους στόχους στην Ευρώπη του 2020 και ήρθε κάποιος από τις επιχειρήσεις από τη Σουηδία και ένας από τους εργαζόμενους και μας είπανε ότι τα διορθωτικά ταμεία έχουν επίπτωση μηδέν. Αυτό μας είπανε. Σίγουρα αυτός ο επιχειρηματίας συγκεκριμένα είχε άδικο να σταματήσει η χρήση των διαθετικών ταμείων. Ωστόσο, δεν είναι σωστό να αφήνουμε τον κόσμο να λένε ότι τα κονδύλια αυτά δεν έχουν θετική επίπτωση. Εμείς με τα νούμερα στα χέρια θα πρέπει να αποδείξουν ότι όντως αποδίδει το σύστημα. Δεν μπορούμε να έχουμε σκόρπιους στόχους από εδώ και από εκεί. Μικρούς διότι αυτό σημαίνει αύξηση του κόστους. Εγώ βρίσκω ότι στη μελέτη αυτή δεν υπάρχει μεγάλο όραμα. Αυτές ήταν οι σκέψεις μου που σας τη λέω ε, μεγαλόφωνα και σας ευχαριστώ για όλα τα στοιχεία που μας Είπα ότι ένας σουηδικός, ε, σουηδός οικονομόλογος δεν ε, ανησυχούσε τόσο για την αποτελεσματικότητα, αλλά είπε ότι τέτοιου είδου κρατικέ ενισχύσει υποσκάπτουν τον ε, θεμητό ανταγωνισμό. Κύριε Γκάφη, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ. Θα ήθελα καταρχήν να πω ότι η αξιολόγηση δεν εστιάστηκε σε θέματα ελέγχου και ήταν εσκεμμένη επιλογή. Πολλοί μας ρώτησαν γιατί δεν ασχοληθήκατε με τον έλεγχο γιατί είπαμε ότι ούτω ή άλλω υπάρχει υπερβολική εστίαση σε αυτά τα θέματα. Εμείς προτιμούσαμε να εστιαστούμε στα αποτελέσματα της ε, πολιτική συνοχής. Να αξιολογήσουμε αυτά τα αποτελέσματα, γιατί υπάρχουν ελεγκτές, υπάρχουν επιθεωρητές. Πάντως τα θέματα της γραφειοκρατίας και του ελέγχου εμφανίστηκαν στην αξιολόγηση. Και διαπιστώσαμε ότι σε ορισμένες χώρες, ιδιαίτερα σε πολλές καινούριες, ξεκίνησε το σύστημα με υπερβολική γραφειοκρατία, αλλά εξελίχθηκε πολύ πιο αποτελεσματικά. Όταν μιλούμε για επιθεωρήσεις και ελέγχους, για να δούμε ποια ήταν τα αποτελέσματα στις περιφέρειες, η προσωπική μου γνώμη ήταν θα ήταν πιο αποτελεσματικό να επικεντρωθούμε περισσότερο στο να προσπαθήσουμε να ενθαρρύνουμε και να παρατρύνουμε τα κρατη να κάνουν περισσότερες αξιολογήσεις των επιτευγμάτων τους στις διάφορες περιφέρειες. Δηλαδή να απομακρυνθούμε από μια προοπτική ελέγχου, όπου μιλούμε μόνο για τον έλεγχο, ότι έχει γίνει κάτι και μετά να επιβάλλουμε κυρώσεις αν δεν έχει γίνει σωστά και να προσπαθήσουμε να απαντήσουμε μια σειρά άλλων ερωτημάτων. Πολλές φορές οι απαντήσεις δεν είναι απλές για τέτοιου είδους αλλαγές που επιδιώκουμε και δεν γνωρίζουμε ότι ένα ευρώ που επενδύσαμε σε συγκεκριμένο τομέα θα έχει απόδοση. Γιατί επειδή είναι διαφορετική κατάσταση της το αποτέλεσμα θα είναι διαφορετικό αυτής της επένδυσης του ενός ευρώ. Και όταν γίνονται αξιολογήσεις, και έχουμε συζητήσεις, υπάρχει λιγότερος φόβος και μεγαλύτερη ειλικρίνεια και εντιμότητα και όλοι μαθαίνουμε αυτή τη διαδικασία και έτσι μπορεί να βελτιωθεί και η ποιότητα των πληροφοριών που δίνονται σε ό,τι αφορά τα αποτελέσματα μιας πολιτικής. Και ίσως πραγματικά έχουμε μια πολιτική διαπαιδαγώγησης, καλύτερης γνώσης, καλύτερης εξοικείωσης, γιατί οι περιφέρειες ενδιαφέρονται ε, για, τις, ε, για την πρόοδό τους, για τα επιτεύγματά τους. Θέλουν να είναι υπεύθυνε γιατί χάραξαν τα σχέδιά τους, αποφάσισαν να δαπανίσουν τα κονδύλια με συγκεκριμένο τρόπο και φοβούνται μερικές φορές την ε, ευθύνη ότι θα πρέπει εμείς να συγκεντρώσουμε τεκμήρια για το κατά πόσο πέτυχαν. Θα προτιμούσα περισσότερη αξιολόγηση να γίνεται στις περιφέρειες και όχι περισσότερη έλεγχη και εξακριβώσεις και αυτό το λέω επειδή εγώ ασχολούμαι περισσότερο με την αξιολόγηση και όχι με τον έλεγχο, καλύτερα να τα αφήσω τα θέματα αυτά στο Γενικό Διευθυντή για να μιλήσει για τη διαφορά αξιολόγηση και του ελέγχου και τι προτιμάτε. Σε ό,τι αφορά τι υπεραπόμακρε περιοχέ, δεν επικεντρωθήκαμε συγκεκριμένα σε αυτές, αλλά από ό,τι ξέρω, αυτή τη στιγμή εκπονείται ειδική μελέτη στην Γενική Διεύθυνση Περιφερειών για τι υπεραπόμακρε περιοχέ. Εμεί δεν μπορούσαμε στην αξιολόγησή μα να τα καλύψουμε όλα, δεν ε, ασχοληθήκαμε με αυτές και από τη συγκεκριμένη αξιολόγηση δεν μπορούν να αντιληφθούν συμπεράσματα για τις υπεραπόμακρες περιοχές, πάντως καταρτίζεται ειδική μελέτη για αυτές. Συμφωνώ απόλυτα μαζί σας ότι τα κράτη-μέλη θα πρέπει να αναλάβουν την ευθύνη και να δείξουν την αποτελεσματικότητα των πολιτικών. Είναι δύσκολο όμως μερικές φορές και δεν υπάρχουν εύκολες απαντήσεις. Και μέσω αυτής της αξιολόγησης και εγώ εντυπωσιάστηκα γιατί ορισμένα πράγματα που ήταν προφανή ότι αν κανείς επενδύσει στις μεταφορές θα έχει οικονομική ανάπτυξη που ήταν λογικό συνειρμός, διαπίστωσα ότι δεν ισχύει. Και μερικοί πανεπιστημιακοί θα μας πούν αυτή είναι η θεωρία. Αλλά στην πράξη τα πράγματα πολλές φορές είναι διαφορετικά. Γιατί έχουμε σημαντικές επενδύσεις στις μεταφορές, για παράδειγμα, που δεν οδήγησαν στην αναμενόμενη ανάπτυξη. Και στο παρελθόν επίσης είπαμε ότι επενδύουμε σε περιβαλλοντική υποδομή για να γίνει μια περιοχή πιο ελκυστική και να δημιουργήσει ανάπτυξη. Αλλά ούτε τέτοιες εμπειρίες είχαμε πάντα. Δεν είναι αυτόματη η σχέση αυτή. Χρειαζόμαστε περισσότερες αποδείξεις, χρειαζόμαστε ανάλυση συγκεκριμένων σχεδίων προγραμμάτων, περιπτώσεων. Θα πρέπει να τα εξετάσουμε όλα αυτά και να δούμε αν πραγματικά υπάρχουν αλλαγές χάρη στην εφαρμογή αυτή τη πολιτική. Πάντω, επαναλαμβάνω, απλέ απαντήσει δεν υπάρχουν. Πάντω, όσο περισσότερε γνώσει συγκεντρώνουμε, και αυτό διαπιστώσαμε με την αξιολόγηση, ότι με την θεματική ταξινόμηση μπορούμε να δούμε τι μα λέει η βιβλιογραφία, τι μα λέει η οικονομική θεωρία και τι γίνεται στην πράξη. Να ελέγξουμε τις διάφορες περιστάσεις, ε, να δούμε τι γίνεται στις διάφορες χώρες, να εντοπίσουμε βέλτιστες πρακτικές και να μεταδώσουμε αυτές τις γνώσεις και μετά να τα συμπηλήσουμε όλα αυτά στη συνοπτική έκθεση. Πάντω σίγουρα πολλά στοιχεία μα μένουν ακόμη άγνωστα και διερεύνητα, αλλά δεν μπορούμε να τα κάνουμε όλα μόνοι μα. Χρειαζόμαστε τη βοήθεια και των περιφερειών και των κρατών μελών. Ο κύριο Άνερ. Θα ήθελα σύντομε παρατηρήσει να κάνω. Καταρχήν, κατά πάσα πιθανότητα θα αντιμετωπίσουμε προβλήματα με την θέσπιση πιο συχνών και συστηματικών ελέγχων. Εγώ πάντως, ε, σε συνεργασία με τους συναδέρφους μου, θα επιδιώξω πιο συχνό διάλογο, πιο ενισχυμένο διάλογο με τις περιφέρειες και οι ε, αξιωματούχοι μας που πηγαίνουν στις περιφέρειες ε, θα προσπαθήσουν να διαμορφώσουν μια καλύτερη γνώμη για το πού λειτουργεί σωστά η πολιτική και πού χωλαίνει. Επίσης κάτι που θα ήταν πολύ σημαντικό φυσικά θα ήταν, όπως είπε και η Βερόνικα, να δημιουργήσουμε μία παιδεία αξιολόγησης. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Και αυτή την παιδεία της αξιολόγησης να την εφησίσουμε και να την μεταλαμπαδεύσουμε στα κράτη-μέλη για να ε, καταλάβουν όλοι ότι όλοι θα βγουν κερδισμένοι από τέτοια εξέταση και γνώση συγκέντρωση γνώσεων στην περιφέρειά τους. Σε αυτό δίνουμε μεγάλη έμφαση. Προσπαθούμε να επιδιώξουμε μια αλλαγή της νοοτροπίας και μια όλο και μεγαλύτερη προσφυγή στις αξιολογήσεις στις περιφέρειες. Και όπως είπε η Βερόνικα, αυτό που είναι πολύ ενδιαφέρον είναι να εξετάζουμε όχι μόνο αμέσως μετά τις περιόδους ε, τον αντίκτυπο, αλλά να εξετάζουμε και τον μακροπρόθεσμο αντίκτυπο συγκεκριμένων σχεδίων και προγραμμάτων. Και έτσι δοκιμαστικά τώρα θα διερευνήσω μία σειρά σχεδίων που έγιναν στην περίοδο 88-93, 94-99, στις πρώιμες φάσεις αυτής της περίοδου, για να δούμε αυτά τα παιδιτικά προγράμματα, πώς απέδωσαν, τι συνέπειες είχαν μέσα σε μια δεκαετία ή δεκαπενταετία. Θα πρέπει να έχουμε μια, μια πιο μακροπρόθεσμη προοπτική. Σε ό,τι αφορά τις υπεραπόμακρες περιοχές, σας ε, διαβεβαιώνω ότι στα πλαίσια της ε, προετοιμασίας μας για την στρατηγική της επόμενης χρονιάς θέλουμε να κάνουμε μία αναθεώρηση και ήδη έχουμε αναθέσει μία σειρά μελετών. Μία από αυτές αφορά τον αντίκτυπο των πολιτικών μας στις υπεραπόμακρες περιοχές και πού η πολιτική μας θεωρείται κατάλληλη για τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους και πού μπορεί να βελτιωθεί. Και ευελπιστώ ότι από τις μελέτες αυτές θα προκύψουν πολύ σημαντικές γνώσεις. Τώρα, το θέμα της απορρόφησης, του ποσοστού απορρόφησης είναι πραγματικά πρόβλημα και θα πρότεινα στους επόμενους μήνες να έχουμε μια δυνατότητα και να σας κάνουμε έστω και μια σύντομη ενημέρωση για το τι γίνεται με την απορρόφηση. Τώρα που έχει περάσει το ίμιση της περίοδου, πάνω από το 70% ή γύρω στο 70% των κονδυλίων δεν έχει ακόμη ε, δρομολογηθεί. Δεν έχει μάλλον προσημειωθεί. Δεν μιλώ για, προ... για πληρωμές, δεν έχει καν ε, αφιερωθεί σε συγκεκριμένα σχέδια. Οπότε θα πρέπει να διαρωτηθούμε τι πήγε στραβά και σε σχέση με τις προηγούμενες περιόδους υστερούμε περίπου ένα χρόνο. Γιατί λοιπόν έχουμε μείνει τόσο πίσω. Γιατί έχουμε μείνει 12 μήνες πίσω. Βέβαια, από ό,τι φαίνεται, όταν ε, παρατείνουμε μία περίοδο για το κλείσιμο της περίοδου του 2006 κατά ένα εξάμηνο και εξαιτία της κρίσης όλα τα κράτη-μέλη έκαναν κάθε προσπάθεια προκειμένου να εκταμιεύσουν και το τελευταίο ευρώ που υπήρχε διαθέσιμο. Και αυτό δημιούργησε συστηματικά μία εξάμεινη καθυστέρηση. Και αναλύουμε και τους άλλους λόγους αυτής της καθυστέρησης σε αυτή την περίοδο. Αλλά θα ήθελα να έχουμε μια ευκαιρία στο μέλλον να έρθουμε και να σας κάνουμε μια παρουσίαση με συγκεκριμένα στοιχεία. Τώρα τι μπορούμε να κάνουμε και τι κάνουμε αυτή τη στιγμή στο συγκεκριμένο τομέα είναι ότι έχουμε όλο και πιο στενές επαφές με τις χώρες και τις περιφέρειες που αντιμετωπίζουν το συγκεκριμένο πρόβλημα, την Ελλάδα Φερρυπίν και η δική σας χώρα κύριε Κυρίλοφ είναι και αυτή που αντιμετωπίζει προβλήματα, αλλά και άλλες περιφέρειες και χώρες αντιμετωπίζουν αντίστοιχες δυσκολίες. Εμείς θέλουμε να προσφέρουμε όλη την αρρωγή και ενίσχυση που μπορούμε στις χώρες αυτές και στις περιφέρειες αυτές για να καταφέρουν να υπερκεράσουν τα προβλήματά τους. Πάντως, πραγματικά είναι σοβαρή ανησυχία αυτή για μας. Σας ευχαριστώ για τις υποδομές των μεταφορών. Δεν είναι επαρκής παράγοντας, δεν μπορεί από μόνο του να δημιουργήσει οικονομική ανάπτυξη, αλλά αν δεν υπάρχει ένας καλός δρόμος, κανένας επενδυτής δεν θα πάει σε μια περιοχή. Χρειάζεται υποδομή για το ελάχιστο επίπεδο προσέλκυσης εθελοντών. Πίτερ Σάιμον. Ευχαριστώ πολύ. Και θέλω να κατασταθέσω ότι πολλές φορές έχουμε στόχους που μπορούν να περιγραφούν ως απλή βελτίωση των συνθήκων διαβίωσης, όπως είδαμε και με τις οδούς και τα λοιπά. Ε, απλώς διότι δεν υπάρχουν επαρκείς τρόποι μέτρησης, αλλά από τους δείκτες που θα χρησιμοποιήσουμε θα πρέπει να δούμε αν είναι ε, δείκτες σχετικοί με την εφαρμογή ή με τα επακόλουθα ενός σχεδίου. Δηλαδή, βελτιώνουμε τι συνθήκε συνθήκες διαβίωσης σε μια περιοχή. Αν φτιάξουμε έναν δρόμο ανάμεσα στο ένα χωριό και το άλλο χωριό, ε, γιατί έτσι επιτρέπουμε στους ανθρώπους να πηγαίνουν πιο εύκολα στη δουλειά τους ε, Και έχουμε πολλές φορές, το έχω δει και εγώ στα σχέδια στην περιοχή μου, ε, αναπάντηχες πολλές φορές ε, συνέπειες, θετικές όμως, ε, θετικό αντικτύπο κάποιων σχεδίων, που επιτρέπει πολλές φορές σε μια περιοχή, παραδείγματι δική μας το είδαμε αυτό, σε μια περιοχή όπου είχαμε σχεδόν γετοποίηση ενός πληθυσμού αλλοδαπών, με την ανάπτυξη μέσω καλύτερων μεταφορών, επαφών με άλλους πληθυσμούς, με ανάπτυξη νέων συνθήκων κοινωνικής συνύπαρξης, κοινωνικού βίου κτλ. Δηλαδή τέτοιου είδους δείκτες νομίζω δεν θα επέτρεπαν ε, να τα, τα γράψουμε αυτά. Στο μπάρι της Απουλίας επίσης που γνωρίζω κάπως καλύτερα ε, πριν από μερικά χρόνια ήταν αδιανόητο κάποιος που δεν ήταν από τον Μπάρι το ίδιο και μάλιστα γέννημα θρέμα του κέντρου της πόλης να μπει μέσα στα τείχη του Μπάρι. Τώρα από την τρομερή εικόνα που μας έδινε πριν από 20-30 χρόνια η πόλη βλέπουμε ότι τώρα έχουμε μια ανθίζουσα, μια άνθηση στην πόλη αυτή, μια ανοιχτή πόλη, μια βελτίωση δηλαδή της ποιότητας ζωής και αυτό είναι κάτι το οποίο σημαίνει ότι ο καθένας μπορεί να πάει όπου θέλει, ότι μπορεί να έχει κοντά του αρκετά ένα λιμάνι, ένα αερολιμένα, ένα δρόμιο, ένα σιδηροδρομική γραμμή. Όλα αυτά νομίζω ακόμα δεν τα έχουμε καν φανταστεί ότι μπορούν να τα επιφέρουν κάποια προγράμματα. Ίσως λοιπόν από την αρχή θα ήταν καλό για κάθε ένα και για κάθε ε, δεκαδικό στοιχείο ενός προγράμματος θα ήταν καλό να έχουμε υπόψη ένα κατάλογο των δυνατόν πλήρη των δικτών που θα ήταν χρήσιμε για να καταγράψουμε τα αποτελέσματα μας προγράμματος. Διαφορετικά πάντα θα αποτυγχάνουμε. Δεν είναι δυνατόν να έχουμε κάποιο μάντι που θα μας λέει τι εξελίξεις μπορεί να φέρει ένα πρόγραμμα από αυτές τις αναπάντηχες όπως σας είπα εξελίξεις ε, εάν προχωρήσει σε υλοποίηση. Πολλές φορές δεν αντα, ε, δεν αντανακλάει πραγματικότητα αυτό το οποίο είχαμε αρχικά υπόψη. Και βέβαια τελικά όλα αυτά, εάν δεν επιτευχθεί ο αρχικά επιδιωχθεί στόχο αλλά κάποιο άλλο, και αν δεν μετρηθεί ο άλλο στόχο βελτίωση των όρων ζωή, τελικά απλώ θα καταγραφεί αυτό το πρόγραμμα σε μια αποτυχία και σε μια διασπάθηση του πόσου χρήματο. Συμφωνώ. Δεν, δεν σας πρόφερα καλά πριν έπρεπε να πω Πέτερ Σίμων. Κάρι Μαντέλ. Σας ευχαριστώ κύριε Άνερα για το ότι επιμείνετε στο λόγο της σχέσης κομισιών και περιφερειών και ξέρω στη Γενική Διεύθυνση ε, ε, θέλετε το προσωπικό να πάει επιτόπου στις περιοχές και σας συγχαίρω γι' αυτό. Έχω πολλές ερωτήσεις. Θα αρχίσω από τους δείκτες όπως τον άφηρε ο κύριος Πίτερ Σιμών. Εισαγωγικά μας είπατε ότι δεν υπάρχουν δείκτες. Ερωτώ, τι δείκτες θα χρησιμοποιήσετε στο μέλλον. Πώς θα μετρήσετε τη βελτίωση του βιωτικού επίπεδου των πολιτών, της ποιότητας ζωής μάλλον, που θα πρέπει να είναι το κύριο μέλημα ε, της πολιτικής. Προς την κυρία Γκαφέ, ξέρω ότι τα αποτελέσματα του Urban θα τα έχουμε μετά από μερικούς μήνες. Ας προδικάσουμε λίγο τα γεγονότα. Μπορείτε να μας πείτε ποια είναι τα κύρια αποτελέσματα της αξιολόγησης του προγράμματος πρωτοβουλίας Urban. Πιστεύω στην Κομισιόν κάποια αξιολόγηση μέσα θα την κάνετε εσωτερικά. Μπορείτε να μου βεβαιώσετε ότι αυτή η κοινωνική πρωτοβουλία ήταν κάτι το θετικό. Αντίθετα το mainstreaming δεν πέτυχε τους στόχους του. Και υπάρχει κάτι που κατεμένει σημαντικό δεδομένων των σημερινών αποτελεσμάτων. Η Κομισιόν θα υποστηρίξει επενδύσεις στις πόλεις και ποια θα είναι η θέση των πόλεων στις επενδύσεις αυτές. Οι πόλεις θα πάρουν άμεσα παραδείγματος κονδύλια του ΦΕΝΤΕΡ. Σαμ Κέλλη. Ευχαριστώ. Θετικά τα αποτελέσματα. Τα περιμένα βέβαια. Δεδομένου των δις που έχουμε εξοδέψει. Δεν είναι περίεργο αυτό. Είπατε στην εισαγωγή σας ότι σας απασχολεί το ότι οι συνάδελφοί σας προβληματίζονται για το πώς δαπανήθηκαν τα χρήματα. Ναι, δαπανήθηκαν, δαπανήθηκαν σοφά. Φρόνημα. Όμως πρέπει να δούμε το διοικητικό κόστος. Μπορεί να μειωθεί. Κόστος εφαρμογής. Και φυσικά το θέμα των απατών που κανένας δεν το δέχεται. Όλα αυτά ως διδάγματα για το μέλλον. Σε μια διεδόδη κατάσταση θα έχετε αυτό που είπε ο κύριος Φανής στο Σίνη. Αλλά αν υπάρχουν κυρώσεις για άτομα που δεν συμμορφώνονται με τις υποχρεώσεις τους, τότε δεν μπορείτε να έχετε εμπιστοσύνη. Γιατί αν δεν υπάρχουν κυρώσεις, αν το ξέρει ο κόσμος δεν υπάρχουν κυρώσεις, θα συμπεριφερθεί με έναν συγκεκριμένο τρόπο. Νομίζω υπάρχει ανάγκη επανεξιολόγησης των περιφερειών και μιλάω για τη χώρα μου όχι τόσο με όρους ε, ΑΕΠ όσο με όρους ε, δυνατότητας δαπάνης. Όσον αφορά την κατασκευή δρόμων, άσχετα με την στρατηγική του 2020, Έχουμε θέματα ανανεώσιμων πηγών ενέργεια, αλλαγή κλίματο. τα οχήματα στου δρόμους, ο αριθμό του θα αυξάνεται συνεχώ τα επόμενα χρόνια, άρα χρειάζονται δρόμοι. Εκεί που δεν έχουν ολοκληρωθεί μεγάλοι αυτοκινητόδρομοι να τελειώσουν. Θα πρέπει όμως να δούμε σε αυτούς που έχουν τελειώσει που υπάρχουν σημεία, μεγάλα σημεία συμφόρησης των οχημάτων. Σε σημεία που τελειώνει ο αυτοκινητόδρομος. Ιδιαίτερα στους ε, ε, δρόμους ε, παρακαμπτήριους γύρω από τις πόλεις. Δακτύλοι κλπ. Αυτά επηρεάζουν την ποιότητα της ζωής, όπως επίσης επηρεάζουν και την κινητικότητα των ατόμων. Και επανέρχομαι σε κάτι που είπα και στην αρχή. Χρειάζομαι μια στρατηγική δημοσίων σχέσεων. Να μπορούν οι πολίτες να δουν ότι όλα αυτά είναι, που προέρχονται από την Ένωση είναι θετικά, έχουν μια θετική επίπτωση στη ζωή τους. Πρόεδρος, έχουμε ακόμα τρεις συναδέλφους με ερωτήσεις πριν ξανάρθουμε πάλι στην Κομισιόν. Η Κομισιόν θα απαντήσει και μετά θα πάμε σε υπόλοιπου τρεις. Η κυρία Κάφρε, η Κομισιόν υπογραμμίζει το πολυπλοκότητα των προγραμμάτων. Το βρήκαμε όλα αυτά στην αξιολόγηση. Όλοι μας θέλουμε αυξημένη δυνατότητα των περιφερειών να τον ορίζουν τα προγράμματά τους να είναι σαφές τι θέλουν να πετύχουν και πώς θα ξέρουν ότι το πέτυχαν ή όχι. Ένα παράδειγμα από την αξιολόγηση του Urban θα σας το πω αμέσως μετά. Πάντα θα γίνονται πράγματα απροσδόκητα κατά κάποιο τρόπο. Αλλά πάντα μπορούμε να βελτιώνουμε την κατάσταση αλλάζοντας τα προγράμματά μας. Και να ξέρουμε κυρίως πότε πετύχαμε στο πρόγραμμα. Οι δείκτες δεν μας λένε τα πάντα. Πολλά γίνονται που δεν είναι δυνατόν να τα συλλάβουν οι δείκτες ναι, να χρησιμοποιούμε δείκτες, αλλά να χρησιμοποιούμε και άλλες μεθόδους αξιολόγησης, συγκεκριμένες μελέτες, case studies, να δούμε τι γίνεται με την πολιτική συνοχή, γιατί πρόκειται για ένα πολύ μεγάλο πλούτο εκεί μέσα. Έχουμε δείκτες σχετικά με οικονομικά θέματα. Έχουμε καλά στοιχεία για το ΑΕΠ, Η δυσκολία είναι ότι δεν παίρνουμε γρήγορα τις πληροφορίες αυτές. Τα τελευταία στοιχεία που έχουμε είναι του 2007. Δεν είναι ιδιαίτερα ικανοποιητικό αυτό. Όταν όμως κοιτάμε θέματα κοινωνικής και γεωγραφικής συνοχής, ακόμα δεν ξέρουμε ποιοι είναι οι σωστοί δείκτες. Και αυτό δεν αφορά μόνο την Ευρώπη. Έχουμε νομπελίστες που προσπαθούν να δουν και να προτείνουν τι δείχτες να προταθούν στο μέλλον που να μετράνε το ε, πώς κινείται η κοινωνία. Ο Στίγκλιτς, παραδείγματος χάρη, το έχει κάνει αυτό. Στην αξιολόγησή μας παίρνουμε στατιστικές εισοδήματο. Να τις χρησιμοποιήσουμε περισσότερο. Αυτές οι στατιστικές και αυτές πάσχουν. Πρέπει να το συζητήσουμε με τις στατιστικές υπηρεσίες, με αυτούς που χαράζουν την πολιτική. Αξιολόγηση για το Urban. Urban. Θα σας δώσω μερικά στοιχεία για την αξιολόγηση ex post. Το αποτέλεσμα είναι γενικά θετικό. Τα προγράμματα Urban ήταν επιτυχή. Έχετε δίκιο όταν λέτε ότι το mainstreaming του Urban δεν έγινε με την έννοια ότι στα τρέχοντα προγράμματα mainstream δεν έχουμε δραστηριότητες Urban. από την άλλη μεριά όμως, μεγάλη δραστηριότητα που υποστηρίζεται από την Urban υποστηρίχθηκαν περίπου στο 60% που είναι μεγάλο νούμερο. Δηλαδή όταν μια δραστηριότητα ξεκίνησε υπό το Urban ένα μεγάλο κομμάτι αυτής της δραστηριότητας αποδείχθηκε θετικό. Και γι' αυτό οι δραστηριότητες αυτές συνεχίζονται με άλλες πηγές χρηματοδότησης στο μέλλον. Τώρα, οι παράγοντες επιτυχίας του Urban είναι πρώτον η εταιρική συμμετοχή, partnership, στόχος μια μικρή περιοχή πιο επιτυχή προγράμματα ήταν αυτά που ε, είχαν σύνδεση με την τοπική αυτοδιοίκηση της πόλης. Αν κάποιος πήγαινε να το κινήσει με, τους, ε, με τον κόσμο γύρω στην πόλη, αν δεν συνεργάστηκε ο Δήμος ή η κοινότητα, η επιτυχία ήταν πιο μικρή. Το Urban είναι ένα παράδειγμα όταν μιλάμε για αξιολόγηση και δείκτες. Στο Urban ήταν και μια χαμένη ευκαιρία. Προσπαθήσαμε εκ των υστέρων να δούμε για τις περιοχές urban που υποστηρίξαμε, να τις συγκρίνουμε με άλλες περιοχές που δεν υποστηρίχτηκαν με την ε, μεθοδολογία αυτή την counterfactual όπως τη λέμε. Δυστυχώς όμως δεν είχαμε τις πληροφορίες και δεν μπορούσαμε να κάνουμε τα ζευγάρια για να γίνει σωστά η σύγκριση. Ωστόσο βρήκαμε ότι πολλές περιοχές αναπτύσσοντα προγράμματα μάζεψαν στατιστικά στοιχεία και πληροφορίες για τα προγράμματα. Η χαμένη ευκαιρία έγκυται στο ότι δεν συνέχισαν περιοδικά να συλλέγουν αυτές τις πληροφορίες σε όλη την περίοδο προγραμματισμού. Αυτό θα ήταν για μας μια καλή πηγή αξιολόγησης της επίπτωσης της πρωτοβουλίας αυτής. Είχαμε ωστόσο παραδείγματα από ένα πρόγραμμα και οι αρχές μάζεψαν πληροφορίες και είπαν ας πούμε ε, θα εξοδεύσουμε τα χρήματα για ανακαίνιση κτηρίων. Ο αξιολογητής είπε όμως ναι δαπανάτε τα χρήματα για την υποδομή αλλά ο αρχικός στόχος ήταν η ανεργία. Πώς έχει, τι επίπτωση γι' αυτό στην ανεργία και δεν ήταν προετοιμασμένοι γι' αυτό. Γι' αυτό πρέπει να είμαστε σαφείς. Τι θα τι θέλουμε να αλλάξει και να έχουμε και μια θεωρία, να έχουμε μια ιδέα κατά νου, αν επενδύσουμε τα χρήματα με τον άλφα τρόπο, πιστεύουμε ότι αυτό, με αυτόν τον τρόπο θα επιφέρει την αλλαγή. Άρα η αξιολόγηση του Urban νομίζω είναι θετική αξιολόγηση. Και όλο και κάτι μπορούμε να διδαχτούμε για το μέλλον. όχι στη δική μου μονάδα, αλλά κάποια άλλη μονάδα έκανε εξολόγηση του διοικητικού κόστους. Το πόρισμα είναι ότι το κόστος δεν είναι τόσο μεγάλο. Όταν ακούμε τον κόσμο που διαμαρτύρεται για τη γραφειοκρατία κλπ. δεν είναι τόσο πολύ αλήθεια αυτό. Για την κατασκευή οδών Αν υπάρχει ένα πρόγραμμα που δεν έχει ολοκληρωθεί, πρέπει να ολοκληρωθεί. Το ερώτημα είναι, θα ολοκληρωθεί με το 2013. Στην περίπτωση αυτή, μήπως θα έπρεπε να επενδύσουμε σε άλλου είδους μεταφορές. Δηλαδή, Μπορεί να μετριαστεί κατά κάποιο τρόπο η υπόθεση ότι ο ρυθμός των οχημάτων θα εξακολουθεί να αυξάνεται αενάως. Οπότε αν δεν έχει ολοκληρωθεί ένας δρόμος, ξέρουμε περιπτώσεις χρησιμοποιήσαμε χρήματα του ΦΕΝΤΕΡ για συντήρηση δρόμων. Για μας αυτό δεν είναι η πιο αποτελεσματική χρήση αυτών των κονδυλίων δίνουμε τα χρήματα να γίνει η υποδομή και μετά να δίνουμε χρήματα για επισκευή ή συντήρηση της υποδομής. Όχι. Αυτό δεν είναι βιώσιμο για μας. Στρατηγική μάρκετινγκ και δημόσιες σχέσεις. Φυσικά υπάρχει περιθώριο βελτίωσης. Στην αξιολόγηση το ενδιαφέρον είναι όταν μιλάμε με τον κόσμο που φιλήθηκαν από τα κονδύλια αυτά. Πολλές φορές μας λένε Πολύ πολύ ενδιαφέρουσες ιστορίες. Ο κόσμος θέλει να μιλάει για τις εμπειρίες αυτές. Και η συλλογή αυτών των ιστοριών είναι πολύ ενδιαφέρον. Φαίνεται πάρα πολύ ενδιαφέρον στοιχείο. Οι περιοχές στόχου 2, όταν οι εξελογητές μιλάνε με άτομα περιοχών τύπου Β, στόχου Β, βλέπουν ότι στην πολιτική συνοχής για αυτούς είναι σημαντικό, τους κάνει να αισθάνονται κομμάτι της Ένωσης, έχει μεγάλη προστιθέμενη αξία, πιο μεγάλη από ό,τι περιμέναμε. Αν χρησιμοποιήσει λοιπόν τα στοιχεία αυτά στο marketing που κάνουμε είτε εμείς είτε εσείς, αυτό θα είναι προς όφελος όλων και της πολιτικής πρώτα και κύρια. Ευχαριστώ πολύ κυρία Βέρντερ και κύριος Μπαφ, παρακαλώ, οι τελευταίο τελευταίοι Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ. Από τόσα είπατε για την παρα... για την παρουσία... με την παρουσία σας παρακολούθησα όσο μπορούσα. Ναι, καλή αξιολόγηση. Αλλά θα ήθελα να μου πείτε εκείνοι οι άνθρωποι, οι περιφέρειες που δεν ζήτησαν χρηματοδότηση έχουν υπολογιστεί, έχουν μπει μέσα στη μελέτη υπήρχαν περιφέρειες που είχαν ανάγκη, θα μπορούσαν να έχουν καταθέσει αίτηση και ενδεχομένως δεν κατέθεσαν. Και γιατί. Ξέρω ότι και εσάς σας απασχολεί ο κύκλος της χρηματοδότησης και ότι δεν υπάρχει επαρκής απορρόφηση των κοντιλίων, αλλά μήπως απλώς δεν είναι αρκετά δημιουργικός ο σχεδιασμός, μήπως δεν υπάρχουν επαρκείς δεξιότητες, στην περιοχή που θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν. Μήπως δεν είναι σε θέση οι ηθήνοντες να προσδιορίσουν ανάγκες. Γιατί βέβαια καλό είναι να κοιτάμε τι δαπανήθηκε και πού, αλλά καλό είναι να βλέπουμε και γιατί κανείς ε, για μια συγκεκριμένη περιοχή δεν εκδήλωσε ενδιαφέρον. Η πρόεδρος, πολύ καλή ερώτηση ασφαλώς, ο κύριος Βλάσικ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Και εγώ πιστεύω ότι άπαξ και ολοκληρωθεί μια συγκεκριμένη περίοδος χρειάζεται για αξιολόγηση. Έχω λοιπόν μια ερώτηση και είναι η εξή. Προφανώς εάν φτιάξουμε μερικά χιλιόμετρα αυτοκινητοδρόμου ή ένα εργοστάσιο καθαρισμού υδάτων και το συνδέσουμε στο δίκτυο κάνουμε κάτι πολύ καλό. Πολύ καλά, μπράβο, όλοι ευχαριστημένοι. Πόσο διαρκεί όμως αυτό το σχέδιο, αυτό το έχουμε καταγράψει, ήταν επαρκής η διάρκεια, η αποδόση του, σχεδίου. Αξιολογήθηκε δηλαδή η αποδοτικότητα των κονδυλίων. Πόσο κόστισε στην Τσεχική Δημοκρατία, την Πολωνία, τη Γαλλία το χιλιόμετρο αυτοκινητοδρόμου που χτίστηκε. Και εν τέλει τα σοβαρότερα προβλήματα που γνώρισε η υλοποίηση του σχεδίου τα καταγράφεται κάπου. Γιατί αυτά βεβαίω θα πρέπει, αυτά πρέπει να δώσουμε έμφαση για να τα αποφύγουμε στο μέλλον. Ευχαριστώ. Ο κύριος Πάφτον, λέει πρόεδρος, με συγχωρείτε, ξεχάστηκα. Μερικά σχόλια. Ίσως την αναφέρθηκαν ήδη βέβαια η απαντήση. Η αξιολόγηση αναφέρει και τα ασθενή σημεία και τον οικονομικό έλεγχο. Ξέρω, το ανάφερε η κυρία Γκάφη, ότι δεν είστε αρμόδιοι για τον έλεγχο. Ωστόσο, αν έχουμε ένα τέτοιο κείμενο, διορθώστε με, νομίζω στήχησε 4,5 εκατομμύρια αυτή η αξιολόγηση, ένα σωρό λεφτά, δημόσια χρήματα, θα πρέπει να υπάρχουν τα νούμερα μέσα σχετικά με τον έλεγχο. Τι ήθελα να μας πείτε πόσα χρήματα δόθηκαν σε πρώτη φάση σε χώρες που ξέρετε ότι δεν έπρεπε να δοθούν λόγω απάτης κλπ. Ή δεν δαπανήθηκαν όπως θα έπρεπε να δαπανηθούν. Πρώτη ερώτηση αυτή. Και δεύτερον, επειδή το, η μελέτη αυτή στήχησε 4,5 εκατομμύρια, δικαιολογείται αυτή τη δαπάνη και θεωρείται ότι έπιασαν τόπο αυτά τα λεφτά. Η κυρία ε, Γκάφη να απαντήσει. Όσον αφορά τι περιφέρειε ή του ανθρώπου που δεν αναζήτησαν χρηματοδότηση, δεν ήταν βέβαια αντικείμενο απευθεία τη μελέτη μα, αλλά προσπαθούμε πάντοτε αυτά τα στοιχεία να τα ενσωματώνουμε στη μεθοδολογία τη αξιολόγηση με την ε, καταγραφή εκείνων που έλαβαν και εκείνων που δεν έλαβαν στήριξη, με την αντιπαράθεση δηλαδή, αυτό που ονομάζουμε counterfactual την αντιπαραβολή. Και βέβαια πρέπει μετά να δούμε με ποια μέθοδο έγινε η επιλογή, με ποια κριτήρια, γιατί κάποιος δεν ε, επέλεξε να κάνει τη σχετική αίτηση. Αυτό μας πρέπει να το δούμε ε, επιπλέον στους συγκεκριμένους τομείς παρέμβασης. Δεν μπορούμε να κάνουμε μια γενικόλογη δηλαδή κρίση για την υπόθεση αυτή. Και καλό θα ήταν και τα κράτη-μέλη να επενδύσουν σε αυτό. για να δούμε αν τα προγράμματα απευθύνονται όντω σε εκείνου που θα έπρεπε να είναι δικαιούχοι του. Και κάτι ακόμη που έχει να κάνει με την επίτευξη των στόχων μακροπρόθεσμα. Γιατί βεβαίω έχουμε ένα πρόγραμμα, ένα στόχο, εξετάζουμε αν τον επιτύχαμε τον στόχο αυτό, αλλά για τις επιδόσεις στοιχεία δεν έχουμε. Μερικές φορές δηλαδή οι στόχοι περιγράφονται ε, κατά τρόπο εσφαλμένα είτε εσκεμένα, γιατί κάποιο θέλει να ορίσει πολύ χαμηλού στόχου για να έχει μετά καλύτερα αποτελέσματα, είτε από ε, άγνοια. Καλό λοιπόν θα ήταν να έχουμε και αυτή τη διάσταση και να προσπαθούμε να την ενσωματώσουμε στην, ε, ε, κατά, κατά την παραβολή μελέτη μας Βεβαίω έχετε δίκιο πιστεύω γιατί και εμείς το βλέπουμε στην αξιολόγηση στην περίοδο 2000-2006 για την Ευρώπη των 10, των 10 τελευταίων των μελών. Έγινε μια προσπάθεια τα χρήματα να αξιοποιούνται σωστά. Ε, μεγάλο επίτευγμα γιατί ήταν οι Κασάνδρες ε, έβλεπαν το αντίθετο. Πλην όμω από την άλλη αυτό σημαίνει και ότι αυξάνεται ο όγκος των χρημάτων 2007-2013 ε, και δεν ξέρουμε αν θα υπάρχει επαρκής ικανότητα απορρόφησης. Ένα στοιχείο που προκύπτει από την αξιολόγηση λοιπόν είναι ότι η πρόταση να διευκολύνουμε περισσότερο τις ανταλλαγές για την ανταλλαγή εμπειριών, τις, τις επαφές για ανταλλαγή εμπειριών εμπειριών και βλέπουμε ότι η επιτυχία στην Ευρώπη ως προς την ε, εφαρμογή στους τομείς πολιτικής θα μπορούσε να αποβεί χρήσιμη. Γιατί να μην προβούμε σε ανταλλαγή απόψεων. Ξέρουμε, Φερρυπίν, ότι η Ισπανία κάνει καλές συνδρομικές γραμμές. Ξέρουμε ότι είναι δύσκολο στην Ανατολική Ευρώπη να προχωρήσουν ε, ε, στο σχεδιασμό αλλά και την εκτέλεση αντίστοιχα προγράμματα συνδρομικά. Γιατί λοιπόν να μην γίνει αυτή η επικοινωνία, γιατί πρέπει να περνάνε αυτά από εμά, από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, γιατί να μην εντοπίσουμε πού υπάρχουν τα δυνατά σημεία στην Ευρώπη, ποιο έχει περισσότερη εμπειρία, καλύτερα αποτελέσματα και να έρθει σε επαφή με εκείνου που έχουν ανάγκη αυτή την εμπειρία. Σε διαπεριφερειακό επίπεδο και μέσα από το Interreg ε, περισσότερο παρά ε, μέσα από θέματα που έχουν πιάνουν μεγαλύτερα κεφάλαια αν θέλετε. Για την αξιολόγηση, πότε και πώς γίνεται. Η απάντηση που θα σα δώσω είναι ότι ακριβώ γι' αυτό λόγο επιλέξαμε 94-99 ε, σχέδια, γιατί θέλαμε να δούμε ακριβώ πώ θα γίνει η αξιολόγηση για την περίοδο 2000-2006. Ναι, μα είπατε εσεί ότι ανήκει στην ε, προϊστορία, αλλά δεν είναι ακριβέ αυτό, γιατί υπάρχουν χώρε οι οποίε ακόμη πάρουν κονδύλια αυτή τη περίοδου 2000-2006 και μάλιστα υπάρχουν χώρε οι οποίε και το 2007 ολόκληρο και το 2008 ολόκληρο είχαν δεσμευμένα κονδύλια και δαπάνες που προέρχονταν από τη χρηματοδότηση του 2000, ε, του 2006. Άρα λοιπόν ε, εκεί που νομίζουμε ότι έχει τελειώσει ένα σχέδιο βλέπουμε ότι τελικά δεν έχει ολοκληρωθεί και όλοι λένε ότι δεν είναι η ώρα να γίνει η αξιολόγησή του. Εγώ στη δουλειά μου κάθε μέρα βλέπω ε, η μισή να μου λένε πολύ νωρίς η αξιολόγηση οι άλλοι μισή, να μου λένε πολύ αργά για αξιολόγηση. Προφανώ ο χρονισμό είναι πολύ δύσκολη υπόθεση. Βεβαίω θα δούμε από τα σχεδια είναι 94-99 ε, κάποιε ιδέε. Ε, ίσως όχι καταληκτικέ, αλλά πάντω αξίζει τον κόπο να επενδύσουμε. Για το κόστος βεβαίως το έχουμε ενσωματώσει. Έχουμε ε, ενσωματώσει το κόστος αναμονάδα των μεγάλων σχεδίων υποδομών όπου καταλήγουμε ότι δεν υπάρχει επαρκή βάση δεδομένων κόστους ανά μονάδα στην Ευρώπη αλλά και πουθενά τον κόσμο με συμπέρασμα και σύσταση ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι σε θέση μοναδική να γνωρίζει και να αξιολογεί αυτό το κόστος και αυτό σημαίνει και επιπλέον βέβαια γνώση του κόστους αναμονάδα και τη δυνατότητα όταν έρχονται νέες προτάσεις για σχέδια να, τα να τις αξιολογούμε, να τις ε, κρίνουμε με βάση αυτή, αυτά τα δεδομένα. Βέβαια και στα κράτη-μέλη μπορεί να αποβεί χρήσιμο το να έχουν τα στοιχεία για το κόστος αναμονάδα. Τα στατιστικά μας είναι περιορισμένα πρέπει να πω, στηρίζονται μόνο στο ΦΕΝΤΕΡ, αλλά πάντως ήταν 96 τα σχέδια 96 σχέδια που ασφαλώς ε, θα έπρεπε να είναι χιλιάδες για να έχουμε επαρκή βάση δεδομένων, αλλά στη βάση δεδομένων θα ενταχθούν σύντομα μέσα από το Ταμείο Συνοχής και τη σχετική αξιολόγηση άλλα περίπου 500 σχέδια και άρα θα έχουμε καλά ε, στέρεα στοιχεία για να προβούμε σε υπολογισμό της μονάδας ε, του κόστους αναμονάδα, του επιδιωκόμενου κόστους αναμονάδα, και της Και βέβαια αυτά δεν τα έχουμε ακόμα και γιατί οι φυσικοί δείκτες δεν είναι συσχετισμένοι με τις κατηγορίες δαπανών. Αυτό θα έπρεπε να το αλλάξουμε στο μέλλον. Θέλουμε άμεσο δηλαδή συσχετισμό μεταξύ του αποτελέσματος και των πόρων που δαπανήθηκαν. Τελευταία ερώτηση. Δεν μπορούμε να αξιολογούμε τα πάντα βεβαίως. Αποφασίζουμε λοιπόν, αφού έγινε αρκετή δουλειά, ελεγκτική, να μην επικεντρωθούμε ιδιαίτερα στην ελεκτική δραστηριότητα κατά την αξιολόγηση, παρότι υπάρχει και ο έλεγχος του δημοσιονομικός μέσα στην ε, ε, αξιολόγηση. Και αφού υπάρχει αυτός ο δημοσιονομικός έλεγχος, μπορούμε να βλέπουμε και ποια κονδύλα θα έπρεπε να έχουν ε, διατεθεί. Ίσως να μην συμφωνείτε εσείς με την ενσωμάτωση εν μέρη του δημοσιονομικού ελέγχου, αλλά πάντως υπάρχει μια λογική που τον, που τον υπαγορεύει. Επίσης έχουμε 16 συμβάσεις αξιολόγησης επιπλέον της ε, συνθετικής πρότασης. Έχουμε πολλές ομάδες δηλαδή αξιολόγηση σε όλη την Ευρώπη, 230 προγράμματα σε όλη την Ευρώπη, προγράμματα διαφορετικών μεγεθών μέχρι 6 δις στο ΦΕΝΤΕΡ, διάφορους τομείς παρέμβασης και υποστήριξη από το ΦΕΝΤΕΡ. Και αυτό που θέλω να πω είναι ότι αποτελεί, πιστεύω, μια καλή απόδοση της επένδυσής μας, διότι έχουμε καλές γνώσεις για δεδομένα, έχουμε στοιχεία για τη χάραξη πολιτικών, πολύ πιο ουσιαστικά από στο παρελθόν. Βέβαια, όπως είπα, γεννά και περισσότερα προβλήματα ακόμη αυτή η αξιολόγηση, αλλά όλο και περισσότερο εστιαζόμαστε, πιστεύω, στην ουσία, δηλαδή να αποδεικνύουμε την ε, αποτελεσματικότητα ή μη Μία πολιτική επιλογής. Και σε αυτό πιστεύω έχει νόημα να επενδύει κανεί. Επίσης ε, η αξιολόγηση και η δαπάνη για την αξιολόγηση. Πιστεύω ότι αξίζει τον κόπο, ιδιαίτερα αν δούμε πόσοι ε, προσπάθεια, πόσο σκόπου έγινε η αξιολόγηση, αλλά και πόσο χρήσιμα στοιχεία προκύπτουν από αυτήν για την Επιτροπή και τα κράτη-μέλη. Το ενδιαφέρον και οι δέσμες βέβαια για την αξιολόγηση έχει ιδιαίτερη σημασία. Θέλουμε δηλαδή να ε, κοινοποιούμε, να γνωστοποιούμε το τι επιτυγχάνουν αυτές οι πολιτικές που αναπτύσσουμε, όχι μόνο για το 2000 με 2006, αλλά ιδιαίτερα με εστίαση στο τι χρειάζεται να αλλάξει ώστε αυτή η πολιτική η περιφερειακή να είναι πιο αποτελεσματική και για το μέλλον. Αυτό νομίζω περισσότερο αποτελεί μια καλή επένδυση. Κύριο Σάνερ, ευχαριστώ. Μου επιτρέπετε δύο στόμες παρατηρήσεις για το ποιος δεν έχει ε, ζητήσει χρηματοδότηση, δεν έχει υποβάλει αίτηση. Να σας πω ότι όντως δεν υπάρχει συστημική μελέτη, αλλά βλέπουμε κάποιον αντίκτυπο απόϊχο αν θέλετε από, τις, ε, από τα στοιχεία αυτά ε, όταν θερυπήν κάποιοι μας επισημαίνουν ότι οι κανόνες είναι υπερβολικά δίσκαμπτοι. Όταν βλέπουμε ότι ενδεχομένως μικρότεροι σκλήμακος δικαιούχοι βρίσκονται σε μειονεκτική θέση. Και αυτό μας επιτρέπει να μελετήσουμε για την προσεχή περίοδο πώς θα μπορούσαμε να αντιμετωπίσουμε αυτό το μειονέκτημα με ενδεχομένως προσεγγίσεις ε, του τύπου καταποκοπήν ποσού, διάθεση καταποκοπήν ποσού, εν πάση περιπτώσει με κάποιο τρόπο να βοηθούμε και τις ε, μικρότερες κλίμακας ε, επιχειρήσεις, τους δικαιούχους μικρότερες κλίμακας, να αξιοποιήσουν αυτά τα σχέδια. Και βλέπουμε ότι υπάρχουν πολλά υψηλής ποιότητα σχέδια, σχέδια στα οποία έχουν ενσωματωθεί όντως νέες και χρήσιμες ιδέες, πίσω από τα οποία ή, μαζί με τα οποία μπορεί να παρουσιάζονται και κάποια άλλα παλαιά και αμφίβολης ποιότητας σχέδια. Θα ήθελα επίσης να πω ότι θα πρέπει κάθε χρόνο να καταμετρείτε το κόστος, να καταμετράτε το κόστος κατά μονάδα και δεν πρέπει καν να περιμένουμε την αξιολόγηση, αλλά συγκεκριμένα κάθε χρόνο να γίνεται αυτή η ε, καταγραφή των στοιχείων. Και βλέπουμε ότι μέχρι το 2008 τα στατιστικά μας δείχνουν πως το ποσοστό σφάλματος τουλάχιστον ως προς την αντίληψη για το ποσοστό σφάλματος ε, από τον πολίτη, από την πολίτη, έχει, είναι αρκετά υψηλό, δηλαδή παρουσιάζει σημαντικό κίνδυνο για την υλοποίηση πολιτικής. Εν πάση περιπτώσει να χτυπήσω ξύλο προς το παρόν δεν ε, θα πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα αισιόδοξοι ω προ την ανάλυση και τα αποτελέσματά τη, δεδομένων και των μεγάλων προσπαθειών στου οποίου έχουμε αποδειθεί από το 2007 μέχρι τώρα και που πιστεύω ότι θα ε, μειώσουν σημαντικά ή θα οδηγήσουν ένα σημαντικά χαμηλότερο ε, ποσοστό σφάλματος. Και όπως είπα, χτυπάω ξύλο γιατί έχουμε μερικές φορές σε σχέση με τις αξιολογήσεις, τώρα να δούμε την αντιπαράθεση των θέσεων μεταξύ κρατών μελών ελεκτικού συνεδρίου και ημών, ε, τώρα κάπου στις αρχές Ιουλίου, για να μελετήσουμε και να διαπιστώσουμε καλύτερα το ποστό φάρματος για το 2009. Αλλά πάνω απ' όλα εδώ πέρα πρέπει να πω ότι κρίνεται η αξιοπιστία της ίδιας πολιτικής μας. Ε, καλά θετικά στοιχεία δεδομένα σε αυτήν την υπόθεση είναι ότι με όλες τις αναλύσεις, με όλες τις έρευνες που έχουν γίνει από τα ευρωπαϊκά μέσα, ε, ελεκτικό συνέδριο, ομάδα πάταξης της ε, ε διαφθοράς, στις τελικές αιτήσει, όταν φτάσει δηλαδή στο τελικό στάδιο η αίτηση, γιατί στην Ευρωπαϊκή Ένωση δηλαδή πλέον, είναι πολύ πιο περιορισμένο το φαινόμενο τη απλή και καθαρής απόπειρα απάτη. Είναι πολύ πιο περιορισμένο. Πλην όμω δεν μπορώ να πω ότι έχει αποτραπεί το φαινόμενο αυτό στο βαθμό που, είναι, που αποτελεί μια γκρίζα ζώνη μεταξύ άγνοια ή αμέλεια και ε, κακής πίστης. Εν πάση περιπτώσει όμως το 6 με 70% Ε, υπάρχουν ε, τέτοιου είδους προβλήματα. Ε, να, να προσθέσω κι εγώ λίγο κάτι για την αξιολόγηση. Γιατί είδατε ότι είμαι ευαίσθητη σε αυτό. Τελειώσαμε δύο συμβόλαια στην αξιολόγηση αυτή. Τα σταματήσαμε σε σχέση με την ποιότητα του έργου της αξιολόγησης. Σας διαβεβαιώνω ότι έχουμε πλήρη επίγνωση του ότι θα ξεδεύουμε χρήματα του Ευρωπαίου Φορολογούμενου για την αξιολόγηση και η αξιολόγηση πρέπει να είναι αποδοτική. Ζητάμε τη μέγιστη δυνατή πληροφορία ό,τι μπορούν να βγάλουν. Σας ε, καθησυχάζω λοιπόν στο σημείο αυτό. Το 2006 είχαμε και το πρόγραμμα του Zoning που επέτρεψε σε ορισμένε χώρε να αποκλείσουν ορισμένου από πρόσβαση στα ταμεία συνοχή. Τώρα το αλλάξαμε από το 2007 και μετά και όλη την επιλέξαμε. Σας ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ για την παρουσίασή σας. Ίσως είστε στην πρωτοπορία σε σχέση με την πολιτική αυτή όσον αφορά την αξιολόγηση. Μην το ξεχνάμε αυτό. Είστε μοναδικοί στην προσπάθεια αυτή αξιολόγησης. Σας ευχαριστούμε και πάλι. Τελειώσαμε τη σημερινή συνεδρίαση της Επιτροπής και θα αρχίσουμε με τη συνεδρίαση των συντονιστών. Αύριο ψηφίζουμε να φέρετε την κάρτα σας. Αμέσως τώρα θα αρχίσει η συνεδρίαση των συντονιστών.